Okay, uh, good afternoon everybody and please... Καλό απόγευμα σε όλους. Ε, σας παρακαλώ καθίστε. Θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα τις ψηφοφορίες. Παρακαλώ καθίστε λοιπόν. Χρειαζόμαστε ησυχία στην αίθουσα. Αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολο για μένα να προεδρεύσω στις ψηφοφορίες. Okay. Uh, on item number two, there is uh, no Ωραία. Λοιπόν, ε, το δεύτερο ε, θέμα στην ημερησία διάταξη είναι έγκριση τη ημερησία διάταξη. Το 3 είναι ανακοινώσει του Πρόεδρου, δεν έχω ανακοινώσει. Τέσσερα, ανακοινώσει ε, του Πρόεδρου σχετικά με τι συστάσει των συντονιστών τη 3η Οκτωβρίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, μπορούμε να θεωρηθούν ότι εγκρίνονται. Το σημείο 5 Δυστυχώ ε, πρέπει να το αναβάλουμε μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, οπότε περνάμε κατευθείαν ε, στο σημείο 6 που είναι η ψηφοφορία για τη διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρωμά. Θα ήθελα να ρωτήσω την εισηγήτρια αν θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. διότι έχουμε πολλές ψηφοφορίε ε, σήμερα εδώ στην αίθουσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδη ε, για τη συνεργασία τους ε, και όχι μόνο αυτού, αλλά και όλους τους συναδέλφου που, συνεισέφεραν στη διαμόρφωση αυτού του κειμένου. Είχαμε πολύ καλέ συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών και υποβλήθηκαν συμβιβαστικέ τροπολογίε με μεγάλη ευκολία. Πολλές νέες καλές ιδέες ε, ε, παρουσιάστηκαν και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, για τη συνεργασία τους πάνω στη γνωμοδότηση και θα ήθελα να πω ότι στον κατάλογο των ψηφοφοριών τα περισσότερα μείων από τη δική μου πλευρά έχουν να κάνουν με επαναλήψει. δεν είναι δηλαδή θέματα τα οποία θα πρέπει να επαρεξετάσουμε. Ε, του είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να κάνω μια παρατήρηση. να βεβαιωθούμε στο μέλλον, ε, να ε, εργαζόμαστε λίγο διαφορετικά. Έχω ε, γράψει και άλλες εκθέσεις για την Επιτροπή μας και στις μελέτες στις οποίες βασίστηκαν οι εκθέσεις ε, διέφερε αρκετά και ε, στην δική μας ε, γνωμοδότηση αυτή λέμε ότι δεν χρειάζονται περισσότερες μελέτες για το θέμα αυτό, δεν χρειάζεται να τα πανούμε χρήματα για περισσότερες μελέτες. Ε, του αντίων ε, είχαμε τέσσερις ε, μελέτες του Κοινοβουλίου στις οποίες στηρίχθηκε η γνωμοδότηση αυτή και ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι οι τρεις από αυτές είναι αμφισβητήσιμες όσον αφορά την, πολιτική, την ποιότητα, η μία είναι αμφισβητήσιμη όσον αφορά την πολιτική ορθότητα και ε, διαβάσαμε το υλικό αυτό ως προετοιμασία στο ταξίδι που κάναμε με την κυρία Μαζόσκα. Ε, Θέλαμε μάλλον να τη διαβάσουμε, αλλά δεν ε, ήταν ε, έτοιμες. Ε, αυτή ήταν η παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους για τη συνεργασία τους και τη συμφορά τους στην έκθεση αυτή, διότι βλέπετε τι γίνεται στην Ευρώπη με του Ρώμα. Κάθε μέρα τα διαβάζουμε αυτά στι Εφημερίδε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μία μη πολιτική, αντικειμενική, αλλά επαγγελματική συζήτηση για το πώ μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση, τι συνθήκε για τι γυναίκε και τα παιδιά αυτά. Ε, δεν θέλουμε μόνο μεγάλε ιδέες από την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο και άλλου ενδιαφερομένους. Θέλουμε δράσει από πλευρά ε, των χωρών και αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα της ε, έκθεσης αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ που με βοηθήσατε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κουρμάη. Θα ήθελα όμως να τονίσω το εξής. Στην σελίδα 3 στον κατάλογο των ψηφοφοριών πριν από τη συμβαστική τροπολογία 12 λέει ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε τις ε, ε, τροπολογίες 62 και 7 της Επιτροπής Απασχόλησης. Δεν θα ψηφίσουμε στο σημείο αυτό αυτές τις ε, τροπολογίες διότι συνδέονται με, την, με τις συμβαστικές τροπολογίες 12 και 15. Μετά λοιπόν την ψηφοφορία της τροπολογίας 15 θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες 62 και 7. Δίνω το λόγο τώρα στην ε, κυρία Γκουρμάη για ένα διαδικαστικό θέμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει όλοι να νιώθουμε κάπως ε, Ρωμά. Ως Ευρωπαία ε, αυτό το μήνυμα ήθελα να στείλω. Αντικαθιστώ την κυρία Κλειβέτη που είναι σκιώδης εισηγητής και δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι παρούσα. Αλλά μετά από τις διαπραγματεύσεις ε, αποφάσισε να στηρίξει τις τροπολογίες σε 36 και 38. Αυτό λοιπόν ε, ήθελα να πω στους ε, συναδέρφους, τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η τροποποίηση. Ας δείξουμε σήμερα ότι είμαστε και εμείς καλοί Ρωμά. Σας ευχαριστώ πολύ και επειδή έχουμε μια πολύ σημαντική κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Αλληλείας. Ε, μας περιμένουν, έχουμε αργήσει. Θα προσπαθήσω να ψηφίσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και εφόσον όταν βλέπω ότι θα υπάρχει σε πλειοψηφία θα ε, προχωράω πιο γρήγορα, αλλά θα διστάζω κιόλα αμέσω μόλι δω ότι δεν υπάρχει σε πλειοψηφία. Σα παρακαλώ λοιπόν σηκώστε τα χέρια σα, ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Ξεκινάμε τι ψηφοφορίε. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές. Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε την 32.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 αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μπορούμε να προχωρήσουμε στη συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε αμέσως. Ελέγχουμε την 54, τροπολογία 54 αρχής πληροφορίας. λήξη της ψηφοφορία. εγκρίνεται. Με μία ψηφο... Το είδα, το είδα. Οι 55 και 56 καταπίπτουν αν έχω καταλάβει καλά. Προχωράμε στη 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε ακόμα την 62 και την 7 της απασχόλησης. Ε, προχωράμε στη συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε την 74 της Επιτροπής Απασχόλησης, λέει ο Πρόεδρος, αλλά λάθος κάνει. 74, Την 74 ψηφίζουμε υπέρ. Ε, ε, συγγνώμη, λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην 76 που είναι προφορική τροπολογία. Υπάρχει καμία αντίρρηση στην υποβολή προφορικής τροπολογίας. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 υπέρ,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 ε, ένα της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δέκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκάξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκαεφτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 της επιτροπής απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Την 33 δεν την ψηφίζουμε, ψηφίζουμε τη συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 είναι προφορική τροπολογία. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει καμιά αντίρρηση στην υποβολή προφορικής τροπολογίας. Είναι ένας βουλευτής κατά. Όχι, όχι, κανείς. Πρέπει όμως να έχουμε δύο αντιρρήσεις ούτως ή άλλως. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 6 ως προφορική ε, τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και έχουμε μια τελευταία προφορική τροπολογία. Υπάρχει καμία αντίρρηση στην υποβολή ε, προφορική τροπολογίας. Όχι. Ωραία, ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίσουμε το σύνολο του ψηφίσματος, αρχή της ψηφοφορίας. And the vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται σαφώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Άννα ε, Ζαπόρσκα που ήρθε μαζί μου πριν από δύο εβδομάδες σε ένα καταβλισμό Ρωμά. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Πολλά μάθαμε. Θα σας τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Και την ε, Κατρίν και την Άντσελα θέλω να τις ευχαριστήσω από τη γραμματεία γιατί ήταν δύσκολη δουλειά που είχαν και βέβαια και τους ε, συναδέλφους μου από το γραφείο μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Άξιζαν τα χειροκροτήματα σίγουρα. Εδώ λοιπόν θα λήξει η Συνδέση Επιτροπή Γυναικών και θα ξεκινήσει η κοινή συνεδρίαση. Σας ζητώ πάρα πολύ συγγνώμη που άργησα. Ζητώ συγγνώμη και στο κρατήριο. Πάντως θα ξεκινήσουμε τώρα την κοινή συνεδρίασή μας με την Επιτροπή Αλίας. Bueno, muy buenas tardes. Καλησπέρα σας. Καταρχά να ζητήσω συγγνώμη γιατί ξεκινάμε με κάποια καθυστέρηση τη δημόσια αυτή ακρόαση. Υπήρχε όμως μια ψηφοφορία όπως είδατε που έπρεπε να προηγηθεί όπως πάντοτε συμβαίνει. Δεν θα καθυστερήσω άλλο λοιπόν. Κυρίσω την έναρξη τη συνεδρίασής μας και καλωσορίζω όλες και όλους ε, εσάς που είστε εδώ παρόντες σε αυτή την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φίλων και της Επιτροπής Αλίας. Καλωσορίζω και χαιρετίζω και τον ε, πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών που κάθεται ξεβονίμων. Ε, είναι πολύ καλό, δεν συνηθίζεται, είναι πολύ καλό να οργανώνονται κοινέ συνεδριάσεις. Αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτή την κοινή δημόσια ακρόαση και για το ετήσιο έργο των δύο επιτροπών του 2013 και είχαμε τρία διαφορετικά πάνελ, όπως ξέρετε. Θα έχουμε μάλλον. Πρώτα απ' όλα να πω δύο σκέψεις, γιατί όσοι με γνωρίζουν θα ξέρουν ότι προσωπικά αποδίδω τεράστια αξία στον ανθρώπινο παράγοντα στην αλία. Πάντοτε θεωρούσα ότι η βιωσιμότητα στην αλία δεν εξαρτάται μόνο από τους ψαρότοπους που θα έχουν πολλά και υγιή ψάρια και γενικότερα θα έχουμε ενδιατήματα υγιή, αλλά και ε, αν υπάρχουν ε, επαρκείς ανθρώπινοι πόροι θα είναι δυνατό κάτι τέτοιο, γιατί οι άνδρες και οι γυναίκες που εργάζονται στην αλία είναι αυτοί που καθιστούν την αλία την αληφτική δραστηριότητα μια αξιοπρεπή εργασία. Πιστεύω ότι είναι άλλωστε και κομμάτι του πολιτισμού πολλών περιοχών και πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Πρέπει λοιπόν να τη διατηρήσουμε και να εξασφαλίσουμε το μέλλον της για τις επόμενες γενιές. Δεν θα σας δώσω στοιχεία αριθμητικά για το πόσο μεγάλη σημασία έχει η παρουσία της γυναίκας στον αλληλευτικό τομέα. Ακόμη και τα επίσημα στοιχεία νομίζω δεν επαρκούν για να καταδείξουν την πολύ μεγάλη σημασία των γυναικών. Αυτό που δείχνουν πάντως τα στοιχεία είναι ότι η γυναίκα διαδραματίζει ζωτικό ρόλο και στον τομέα της αλληλείας και έχουμε πολύ μεγάλα παραδείγματα ε, γυναικών ε, που πολλούν ε, ψάρια ή που επιδιορθώνουν δίχτυα ή που εργάζονται σε άλλες τομείς της αλληλευτικής δραστηριότητας και πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές φορές ε, παίρνουν και τη θέση του συζύγου τους όταν αυτός βρίσκεται στα ανοιχτά πάνω στο αλληλευτικό σκάφος. Τα δικαιώματα και των γυναικών αυτών δεν έχουν αναγνωριστεί απόλυτα. Πρόοδος έχει σημειωθεί μεγάλη, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και ένα σημαντικό κομμάτι των προκλήσεων ε, θα το αντιμετωπίσουμε, αν θέλετε, και με τη σημερινή ακρόαση. που είμαι βέβαιος ότι θα διδαχθούμε όλοι πολλά από αυτήν την ακρόαση. Πριν ξεκινήσουμε, να πω ότι θα συμπροεδρεύσουμε οι δύο πρόεδροι, ο συνάδελφος Μικάλη Γκούσταυσον και εγώ της συνεδρίασης αυτής. Θα δώσω το λόγο στην πρώτη ομιλήτρια, που καλωσορίζουμε είναι η Γενική Διευθύντρια Ναυτικών Υποθέσεων, Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλίας είναι η κυρία Λόρι Εύμας που θα μας δώσει ε, την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν ακούσουμε όμως την κυρία Εύμας θα δώσω το λόγο για να χαιρετισμό στον κύριο Γκούσταυσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να χάσουμε χρόνο διότι καθυστερήσαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μάτο και την Επιτροπή Αλίας για την κοινή αυτή συνεδρίαση. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό και ξέρω ότι η ε, Επιτροπή σας ε, λαμβάνει υπόψη τα θέματα ισότητας. Ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ λοιπόν που έχουμε αυτήν την κοινή ακρόαση και καλό θα είναι να έχουμε και μια κοινή έκθεση από όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λόρι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ του αφεντικού μου. Θα ήθελε να είναι εδώ ε, αλλά δεν τα κατάφερε οπότε είμαι εγώ η τυχερή. Οι συμπρόεδροι Μίκαλ και Γκάμπριελ πολύ σωστά έλαβαν, ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία. Είναι πολύ επίκαιρη. εξαίρετο timing. Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες στην Αλία ήδη συνεισφέρουν πολλά. Πιστεύουμε όμως ότι μπορούν να συνεισφέρουν ακόμα περισσότερα. Η πρόταση την οποία συζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας αναγνωρίζει ρητά το ρόλο των γυναικών στις κοινότητες αλίων. Στόχος για το μέλλον είναι να διευκολυνθούν και να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στο ε, δυναμικό των γυναικών. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή για το μέλλον από ό,τι δείχνουμε σήμερα. Ποιο είναι το πλαίσιο. Το οικονομικό πλαίσιο ε, αποτελεί μια πρόκληση και για αυτό το τομέα. Και ποια είναι η πρόκληση, η δημιουργία περισσότερης απασχόλησης και ανάπτυξης. Και εδώ, όπως και στους άλλους τομείς οικονομίας και το νέο χρηματοδοτικό μέσο θα πρέπει να μας επιτρέψει να το κάνουμε αυτό. Από πού ξεκινάμε. Κοιτώντας το θέμα του πλευρά των γυναικών. Οι γυναίκες παίζουν ήδη σημαντικό ρόλο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 100.000 γυναίκες που ξεκιναμε κοιτωντας το θεμα του πλατών των γυναικων οι γυναικες παιζουν ηδη σημαντικο ρολο στην ευρωπαικη ενωση εχουμε 100000 γυναικες που απασχολουνται στον τομέα της αλίας. Πάνω από το 25% δηλαδή του συνόλου των απασχολούμενων στον τομέα. Αν ε, δούμε όμως ε, λίγο πιο λεπτομερό το θέμα θα ανακαλύψουμε ότι μόνο το 4% των αλλιέων είναι γυναίκες. Στην ηχθειοκαλλιέργεια οι γυναίκες είναι ανεβαίνουν στο 30% και αν δούμε στη, τη μεταποίηση εκεί οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του εργατικού δυναμικού. Και ε, πολλά κρύβονται πίσω από αυτήν την κατανομή. Ε, Γκαβριέλ, ε, συμμετείχα στο τρίτο συνέδριο των γυναικών στην Αλία, στο Σαντιάγο, στη Χιχόν μάλλον. Ε, και εκεί είδαμε τα καλύτερα παραδείγματα δικτύωση των γυναικών σε όλη την Ευρώπη. Εκεί πάλι συζητήσαμε το θέμα των κρυφών γυναικών. Το, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει αναφέρει. Τι είναι αυτές οι κρυφές, οι κρυμμένες γυναίκες. Πρώτον, και πάνω απ' όλα σημαίνει ότι πολλές γυναίκες δεν καταγράφονται στις στατιστικές διότι εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις ε, δεν απασχολούνται όμως επισήμως, ε, ε, δεν είναι ασφαλισμένες και ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλές γυναίκες όπως γυναίκες που συλλέγουν μαλάκια ή επιδιορθώνουν δίχτυα που εργάζονται σε πολύ επισφαλείς συνθήκες. Δεύτερον, τι άλλο δεν δείχνουν τα νούμερα. Δεν δείχνουν το γεγονός ότι πολύ συχνά οι γυναίκες έχουν εργασίες ανειδίκευτου εργάτη ε, και δεν έχουν πολλές δυνατότητες εξέλιξης. Η άλλη διάσταση που δεν δείχνει τα νούμερα είναι η κοινωνικο-οικονομική συνεισφορά των γυναικών στις τοπικές κοινότητες, πέραν δηλαδή της εργασίας τους. Μιλάμε για την ανθρώπινη διάσταση, για την οποία μίλησε και ο Γκαβριέλ. Θα πρέπει να είμαστε, ε, ε, να είμαστε ε, να αντιληφθούμε το που βρισκόμαστε σήμερα, αλλά θα πρέπει να αντλήσουμε και εμπειρία και έμπνευση από το παρελθόν. Κάτι πολύ θετικό είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας έχει δώσει στις γυναίκες τη δυνατότητα να αναζητήσουν καινούργιες ή πρόσθετες πηγές εισοδήματος και να συνεισφέρουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κοινωνιών τους. Το ίδιο θα κάνουμε και με το καινούριο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Το νέο αυτό ευρωπαϊκό πλαίσιο θάλασσας και αλλιά θα δίνει στις γυναίκες τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε κατάρτιση, ε, να δημιουργούν δίκτυα για να ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά κυρίως το Ταμείο αναγνωρίζει ρητά όχι μόνο τις αλληλείς γυναίκες, που δεν είναι και πολλέ, αλλά και συζύγους και συντρόφους αλλιέων. Οπότε και αυτές μπορούν άμεσα και ατομικά για πρώτη φορά να είναι δικαιούχοι χρηματοδότησης. Για παράδειγμα για τη βελτίωση ε, των προσόντων ε, διαχείρισης και ε, ή τη δυνατότητα χρηματοδότησης προς, ανάπτυξη προσόντων για να γίνουν πιο κερδοφόρες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βοηθήσουμε ταυτόχρονα και τις κοινότητες και τις επιχειρήσεις να αντλήσουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση, να αυξήσουν την προσθέμενη αξία των προϊόντων τους και το σημαντικό είναι να υποστηριχθεί η, ε, η δραστηριότητα στη στεριά, δηλαδή η μεταπίεση και η εμπορία. Εκεί ήδη κάνουν πολλά γυναίκες και μπορούν να κάνουν και περισσότερα στο μέλλον. Επίσης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες θα παίξουν πιο σημαντικό ρόλο στην, στα προγράμματα εφαρμογής που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της θέλει να ενισχύσει την, την ε, διάσταση του φύλου Οπότε στη νέα προγραμματική περίοδο, από το 2014 και μετά, οι γυναίκε και ενό γυναικών θα μπορούμε να μένουμε ότι θα παίξουν ένα σημαντικότερο ρόλο και κατά τη φάση του προγραμματισμού. Θα πρέπει δηλαδή να του ζητείτε γνώμη τη στιγμή που ε, επεξεργάζομαστε τα προγράμματα και θα υπάρχουν μέτρα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή του στα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα. Αυτό θα ληφθεί υπόψη από την αρχή, από την διαδικασία επιλογή. Βέβαια, οι γυναίκε θα πρέπει να συμμετάσχουν και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων εν τη εξέλιξη του. Είναι λίγο γραφειοκρατικό, αλλά θα είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί ξέρουμε ότι οι γυναίκε ω τώρα δεν συμμετέχουν επαρκώ. Πέραν αυτή τη ε, διαρθρωτική και διοικητική αλλαγή θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επίση ότι τα, θα λειτουργήσουν τα μέτρα δικτύωση και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Ε, μεταξύ αυτών και βέλτιστων πρακτικών στην ε, ε, ισότητα των δύο φύλων. Επίσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποβάλουν επαρκείς αναφορές και στοιχεία έτσι ώστε και εμείς και το Κοινοβούλιο να μπορούμε να παρακολουθήσουμε από κοντά την όλη διαδικασία. Συνοψίζοντας να σας πω το εξής. Ο, ο γενικότερος στόχος ε, είναι να δώσουμε στις γυναίκες καινούριε δυνατότητες και να βελτιώσουν τις δικές τους ε, δυνατότητες ε, πρόσληψης αλλά και αυτές της οικογένειάς τους και των τοπικών τους κοινωνιών. Αυτή η συζήτηση λοιπόν γίνεται στην βέλτιστη δυνατή στιγμή στη διαδικασία, στην νομοθετική διαδικασία γιατί ε, αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο έχει κοιτάξει την πρόταση κομισιών ε, και θα ξεκινήσει λίγο τριμερή τριμερής Έχουμε κάποια πρώτα διδάγματα, ε, έχουμε κάποιες θετικές εμπειρίες πάνω στις οποίες θα χτίσουμε, θα οικοδομήσουμε και ελπίζω ότι θα ακούσουμε και καινούριες ιδέες σήμερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Evans. Θα περάσουμε λοιπόν τώρα χωρίς καθυστέρηση στα τρία πάνελ. Το πρώτο με θέμα τις γυναίκες ε, στην Ευρωπαϊκή Αλία και Θεοκαλλιέργεια, σημερινή κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές. Πριν ακούσουμε τι παρουσιάσει όμω. θα ήθελα να δώσω καταρχά το λόγο στην Ντολόρε Γκαρθία Ιέρο, η οποία είναι η συντάκτρια μια έκθεση ίδια πρωτοβουλία, είναι μέλος επιτροπή Αλία. Θα μα κάνει λοιπόν την εισαγωγή και εν συνεχεία θα δώσω το λόγο στο Ραούλ Ρομέβα, που είναι συνεισηγητής ε, μέλο επιτροπή ε, για τα δικαιώματα τη γυναίκα και τη ισότητα φίλων και ο Ραούλ είναι μέλος της Επιτροπής Αλίας όμως, οπότε γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση. Και μετά τις δύο αυτές παρεμβάσεις θα περάσουμε ευθύ αμέσως στα υπόλοιπα μέλη του πάνελ. Δολόρες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών, κυρίες και κύριοι, τεχνική οργανώσεις ε, των πολιτών, ε, γυναικείες οργανώσεις, όλους θέλω να σας ε, καλωσορίσω και πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας αυτή. Η έκθεση πρωτοβουλίας, σε οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος Επιτροπής Αλίας, αποτελεί καρπό δουλειάς που κράτησε πάνω από ένα χώρο. Και εδώ, χρόνο και θέλω εδώ να ευχαριστήσω γιατί είχα την υποστήριξη της Επιτροπής. Ήταν πολύ δύσκολο, έπρεπε να μελετήσω τις προτάσεις και των ε, τεσσάρων κανονισμών αλλά και τις εκθέσεις που συζητήθηκαν ε, μέσα σε αυτή τη χρονιά και θα έπρεπε βέβαια να καταθέσουμε και τροπολογίες. Οι τροπολογίες αυτές έχουν ενσωματωθεί πλέον και είναι πολύ ε, σημαντικές γιατί θέλουμε να υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και στον τομέα της αλίας και της χθεκαλλιέργειας και χαίρομαι πολύ γιατί είναι κοινή έκθεση, έκθεση της Επιτροπής Αλίας και της Επιτροπής ε, για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Και έτσι εμπλουτίζεται ακόμη περισσότερο ο στόχος που είχαμε στη δική μας Επιτροπή. Δηλαδή θέλουμε και τις οικονομικές και τις κοινωνικές συνθήκες ε, των γυναικών να τις βελτιώσουμε. Πολλές φορές με την αφανή τους δουλειά που δεν αναγνωρίζεται σε πολλές οικογένειες, σε πολλές περιφέρειες, όπως είναι ακόμη η Γαλλικία, ε, καταφέρνουν να επιβιώνουν, ιδίως αυτές τις δύσκολες στιγμές ε, της κρίσης της οικονομικής που βιώνουμε όλοι. Θέλω επίσης να πω ότι το 2005 και το 2010 προκάτοχοί μου έκαναν κοινή πρόταση για την λήψη μέτρων και αυτά τα μέτρα τα επαναλαμβάνω και εγώ. Κοινή οργάνωση αλίας, Ευρωπαϊκή Οργάνωση Αλίας, εξωτερική πολιτική, το Ταμείο για την Αθλητική Θάλασσα που συζητάμε και αυτή η έκθεση, όλα αυτά για το ρόλο των γυναικών, για την κρίση κλίμακα παράκτη αλία. έγιναν ε, πράξη χάρη στην ε, συμμετοχή όλων των βουλευτών. Και σε αυτά τα κείμενα δεν αναφέρονται ε, απλά οι στόχοι, αλλά υπάρχει υποχρέωση από πλευρά Κομισιόν να κάνει πράξη όλα αυτά. Τα 12% των γυναικών ε, συνολικά εργάζονται στον τομέα της αλληλείας με βάση τα επίσημα στοιχεία, της, επίσημες στατιστικές ε, που συγκεντρώνονται αναφύλλω, διότι αν διαβάσουμε προσεκτικά και αναζητήσουμε δεδομένα όπως κάναμε εμείς όλο αυτό τον καιρό, και θα παρουσιαστεί σήμερα μια μελέτη, θα δούμε ότι το ποσοστό αυτό είναι πιο μεγάλο. Ανέρχεται στο 14% και 16% ε, η γυναικεία αυτή η παρουσία σε αυτές τις δραστηριότητες. Γι' αυτό τις λέμε κρυφή ε, την παρουσία αυτών των γυναικών. Και θα πρέπει πάρα πολύ ε, να τονίσουμε και να προβάλλουμε το ρόλο των γυναικών και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. σε κάθε επίπεδο από πλευρά ιδίω των ε, αρμόδιων αρχών. Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών ε, από το 2015 στο 2020 θα ισχύει και αυτός είναι ένας από τους στόχους της στρατηγικής αυτής. Θέλουμε να μην υπάρχει επίση διακριτική μεταχείριση στον τομέα των μισθών, επαγγελματικά και ούτω καθεξή επίση η κατάρτιση, επαγγελματική εκπαίδευση και ε, γέννη η εκπαίδευση των ε, γυναικών και ιδίω των νέων σε όλα τα επίπεδα, στα συνδικάτα, στις αλευτικές οργανώσεις, ε, στη, στα τεχνικά κλιμάκια, στη διαχείριση είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί θα βοηθήσει να ε, περάσει η σκητάλη και στην επόμενη γενιά, σε επόμενες γενιές, ιδίως για τη μικρή παρακτία αλία και ιδίως για τις περιφέρειες που κυρίως ε, ζουν από αυτή τη δραστηριότητα. Επίσης θα πρέπει να εγγυηθούμε την ισότητα και την μισθολογική, την ισότητα μισθολογική μεταχείριση, την νομική προστασία, την προστασία την υγειονομική, την οικονομική επίσης ενίσχυση όταν ε, μια γυναίκα δεν μπορεί να εργαστεί για βιολογικούς λόγους, για κάποιο ε, φυσικό, φυσική καταστροφή, για κάποιο άλλο λόγο. Ε, και αυτά θα τα δούμε, θα συζητήσουμε και το Οικονομικό και Ναυτικό Ευρωπαϊκό Φόρουμ και με τα συμβουλευτικά όργανα και με τα όργανα λήψη αποφάσεων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να έχουμε διαβουλεύσει, πρέπει να ενισχύσουμε την συμμετοχή και πρέπει να στηρίξουμε τι ενώσει των γυναικών, τα συμβουλευτικά όργανα με διάφορα project συγκεκριμένα. Όσοι οι Ισπανοί ε, πραγματικά νιώθω υπερήφανοι γιατί η χώρα μου κάνει αυτά που λέω και είμαστε απόδειξη τότε όταν υπάρχει θεσμική στήριξη μπορούμε οι γυναίκες να οργανωθούμε και να ε, βοηθήσουμε τον ε, τομέα αυτό, ιδίως ε, μια, ένα κλάδο πολύ ευαίσθητο που είναι η ηλεκτρία σωστράκων. Πρέπει όλα αυτά να ληφθούν ε, υπόψη και πρέπει όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέρει και η Διεθνής Οργάνωση να γίνουν πράξη. Πολιτική συμμετοχής, δικαιώματα ανδρών και γυναικών, Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη και να λαμβάνονται και όταν υπογράφονται πρωτόκολλα στι με χώρε. Επίσης πρέπει να αναφέρω πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προβλήματα υγείας. Επειδή είμαστε σε πάρα πολύ, μιλάμε για ένα, μια δουλειά πάρα πολύ ιδιαίτερη, είναι θέματα τα οποία χρήζουν απάντησης και πρέπει να τα δούμε άμεσα, ιδίως για τις ε, γυναίκες που διαπληρώνουν δίχτυα, για τις ε, συλλέκτριες οστράκων, που πραγματικά πολλές από αυτές ε, υποφέρουν προβλήματα υγείας. Πολύ συγκεκριμένα. Τέλος, πρέπει αυτό το ψήφισμα της 10 Σεπτεμβρίου του 2012 του Κοινοβουλίου μας να εξασφαλίσει ότι εν γέννη η νομική, η κοινωνική αναγνώριση και η καλύτερη ανταμοιβή ε, των γυναικών για το ρόλο που διαδραματίζουν στον ελευτικό τομέα να γίνει πραγματικότητα. Να έχουν τα ίδια δικαιώματα άντρες και γυναίκες και να έχουν και συγκεκριμένο νομικό καθεστώς ε, και κοινωνικά επιδόματα ίδια με αυτά που έχουν οι, ε, που έχουν οι ανεξάρτητοι επαγγελματίε και οι σύντροφοί τους ή συντρό... άντρε άντρες και ανάλογα. Θέλω να σα ευχαριστήσω όλου. Θα έχουμε τη δυνατότητα άπαξ και κατατεθεί επίσημα η έκθεση αυτή πρωτοβουλία να τα συζητήσουμε όλα αυτά σε μεγαλύτερο βάθο και φαντάζομαι ότι θα μπορέσετε κι εσεί να μα δώσετε τι δικέ σα ιδέε για να εμπλουτίσουμε και να βελτιώσουμε το κείμενο. Ολοκληρώνοντα, θέλω να πω ότι πραγματικά το κάθε ειλικρίνεια ε, αποτελούν για μένα μεγάλο προνόμιο γιατί είχα από την αρχή τη στήριξη όχι μόνο τη δική μου πολιτική ομάδα, αλλά και του Προέδρου τη Επιτροπή μα, τη Επιτροπή Αλία. Και έτσι κατάφερα ολοκληρώσω αυτό το έργο. Σα ευχαριστώ πολύ. Πρώτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δολόρες, τώρα θα δώσω το λόγο στον Ραούλ Ρομέβα. Θα είμαι σύντομο. συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε η Ντολόρε Γαρθία Γέρο και ταυτόχρονα εκτιμώ ιδιαίτερα τόσο τη δική της δουλειά όσο και άλλων συναδέλφων. Αυτό εδώ σήμερα είναι ένα ε, ακόμα βήμα που συμπίπτει και με τις συζητήσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσας και Αλίας. Ε, εγώ είμαι μέλος και των δύο επιτροπών που συνσυνεδριάζουν σήμερα, οπότε ε, έχω και τις δύο οπτικές. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το βασικό θέμα ουσίας, το οποίο είναι η αφάνεια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τις καλεσμένες μας, ε, τις οποίες και έχουμε προσκαλέσει ακριβώς για αυτό το λόγο. Θα σας δώσω το λόγο και θα επιστρέψουμε ερωτήσεις ενδεχομένω. Ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα, λέει ο Πρόεδρος. Περνάμε στους εμπειρογνώμονες που έχουμε καλέσει. Ο λόγος καταρχήν στην, κυρία, στην Κάτια Φραγκούδη, ε, Πανεπιστήμιο της ε, Βρέστης. Η γυναίκα στην Αλία, Ευρωπαϊκή Προοπτική, είναι ο τίτλος του θέματός της. Ε, της δίνουμε το λόγο. Μανέρα resumida, evidentemente. Señora Francrudes, tiene la, la palabra. Bonjour. Euh, Καλή σας μέρα. Για δεύτερη φορά έχω την χαρά να απευθυνθώ ε, σε μέλη του Κοινοβουλίου. Πρώτη φορά ήταν το 2008, τώρα πέντε χρόνια μετά να δούμε τι έχει αλλάξει. Σα ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο όργανο το οποίο έχει εκδώσει δύο εκθέσεις, ε, εξεραστεί δύο εκθέσεις για το ρόλο των γυναικών στην Αλία, στον τομέα της Αλία. Η έκθεση αυτή ε, που σας παρουσιάζω ε, μελετά τέσσερα θέματα. Το θέμα των στατιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα και η σημασία τους για την αναγνώριση των γυναικών και του ρόλου τους. Δεύτερον, ο ρόλος των συντρόφων και συζύγων, των αλίων, τους οποίους ε, βοηθούν και συνεισφέροντας και, και στην οικογενειακή οικονομία. Τρίτον, τα δίκτυα των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού βρισκόμαστε, ποια είναι η σημερινή κατάσταση, τι έχει επιτευχθεί από το 2008 και μετά. Και κατόπιν, επίσης να πω ότι τι άλλο, τι χάσαμε επίσης από το 2008 και μετά, γιατί δεν έχουμε κερδίσει μόνο. Και τέλος, λέω, ο ρόλος των ε, γυναικών ε, στην ε, κοινή αλληλευτική πολιτική. Καταρχήν, ήμουν λίγο σκεπτικιστική σε ό,τι αφορά, διστακτική σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, γιατί το 2008 δεν είχαμε και πολλά στατιστικά στοιχεία. Ε, δεν ήταν εύκολο να δούμε πόσε ήταν οι γυναίκε που εργάζονταν στον τομέα τη αλληλεία εκείνη την εποχή. Όπω ε, βλέπετε, καταρχήν παρουσιάζω τα στατιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο, τα παγκόσμια στατιστικά, 45 εκατομμύρια άτομα, άνδρες και γυναίκε που εργάζονται στην Αλία, σύμφωνα με τον ΦΑΟ, 12% του εργατικού δυναμικού το 2008 ήταν γυναίκες. Ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντίθετα με τα όσα ελέγχθηκαν προηγουμένως, 12,6% του συνόλου του εργατικού δυναμικού της Αλίας είναι γυναίκες. Ήταν γυναίκες το 2012. Ε, αφορά κυρίως τη μεταποίηση, την αλία και την ηθιοκαλλιέργεια. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από την Eurostat. Η Eurostat δίνει στατιστικά για ένα αριθμό χωρών, όχι για όλες τις χώρες. Προς το παρόν απλώς παρουσιάζω τα στατιστικά στοιχεία, θα τα κρίνω αργότερα. Από το 2008 και μετά ε, έχουμε και ε, πλέον ε, στοιχεία, στατιστικά στοιχεία με ρητή αναφορά σε άνδρες και γυναίκες. Το 28% ε, του εργατικού δυναμικού στην ηχθειοκαλλιέργεια είναι γυναίκες και το 56,6% του εργατικού δυναμικού που δουλεύει, που εργάζεται στη μεταποίηση είναι επίσης γυναίκες. Αντίθετα όμως για τους αλληλείς δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία. Γιατί, Γιατί ε, η αναφύλλο κατανομή είναι υποχρεωτική ε, μόνο για τη μεταποίηση και τις ηχθειοκαλλιέργειες, όχι όμως και για την αλλία. Εδώ θα δείτε τα στατιστικά στοιχεία διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, όπως τα δίνει η Eurostat. Βλέπετε υπάρχουν κράτη-μέλη που δίνουν στοιχεία και υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν παρέχουν τέτοια στοιχεία. Ε, δεν είναι υποχρεωμένες οι χώρες να κάνουν την κατανομή μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα και όταν την κάνουν, ε, το σύνολο ε, είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των ανδρών. Οπότε τι το ερώτημα αν το, η διαφορά είναι οι γυναίκες. Ε, αν δούμε τα στοιχεία του Eurostat είναι αυτά, ενώ αν τα, συγκρίνουμε με τις ΤΕΣΠΗ, βλέπουμε ότι το 3% ε, είναι γυναίκες, 32% ε, μάλλον στην αλία, το 32% στην Χθιοκαλλιέργεια και το 65% στην μεταποίηση. Είναι ο συνδυασμός των δύο στατιστικών πηγών που δίνει αυτά τα αποτελέσματα. Υπάρχει λοιπόν μια ε, διαφορά, μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα διάφορα στατιστικά στοιχεία που λαμβάνουμε. Ε, δεύτερον, έχουμε στατιστικά μόνο για 14 κρατημέλη. Και όπως έλεγα προηγουμένως, το σύνολο της, των, του εργατικού δυναμικού ε, είναι μεγαλύτερο από τη, τις θέσεις εργασίας των γυναικών, οπότε θεωρούμε ότι το, η διαφορά είναι οι γυναίκες. Από την STCF ε, έχουμε πλέον στατιστικά στοιχεία γυναίκες και άντρες χωριστά, αλλά μόνο για την ηχθειοκαλλιέργεια και τη μεταποίηση, όχι μόνο για την αλία. Άλλωστε μόνο 16 κρατημέλη έδωσαν στατιστικά στοιχεία, 4 κρατημέλη δεν έδωσαν κανένα στατιστικό στοιχείο και 2 κρατημέλη ε, μας έδωσαν στοιχεία μόνο για τους άνδρες. Αυτά σε ό,τι αφορά τα στατιστικά που έχουμε το 2013 στην Ευρώπη. Μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, είναι σαφές, και ίσως το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας μπορεί πράγματι να χρηματοδοτήσει, ε, μάλλον να καταστήσει υποχρεωτική την κατανομή των στατιστικών στοιχείων ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών, να να γίνει υποχρεωτικό να ληφθούν υπόψη και άλλοι δείκτες κλπ. Αυτή τη στιγμή ο μόνο κοινωνικό δείκτης ε, τη Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλία είναι η απασχόληση. Ακόμα και έτσι όμω, τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι εξαιρετικά. Οπότε τίθετο ερώτημα ακόμα και για το κατά πόσο λειτουργεί αυτό ο δείκτης που είναι ο βασικό δείκτη τη ε, κοινή ε, πολιτική Αλία. Τώρα, περνάμε στην αμφάνεια, σε αυτό που ονομάζουμε αφάνεια, στις ε, συντρόφους ε, και στις ε, βοηθούς ή τις συζύγους σε αλληλευτικές επιχειρήσεις. Γενικά πρόκειται για εργασία μη αμοιβόμενη, μη δηλούμενη, αδήλωτη εργασία συνήθως. Οι γυναίκες αναλαμβάνουν πολλά παραδοσιακά καθήκοντα, διοικητικά, αλλά και άλλα που έχουν σχέση με τη στεριά, τις επαφές με την εθνική διοίκηση, τους, τα σωματεία των ε, αλλιέων, ε, με τις τράπεζες κλπ. Πολλές φορές πολλούν ψάρια οι γυναίκες ε, στην αγορά ή σε άλλα σημεία. Ε, πολύ συχνά επίσης καθαρίζουν τα όστρακα, ε, τα πακετάρουν, τα συσκευάζουν και πρόσφατα, τελευταία, τους έχει δοθεί και το καθήκον της διαφοροποίησης. λέει δεδομένου ότι τα εισοδήματα από την Αλία δεν είναι αρκετά, οι γυναίκες υποχρεώνονται να αναπτύξουν και ε, καινούργιες δραστηριότητες εργάζονται σε μικρές μεταπτυχικές επιχειρήσεις, ε, σε εστιατόρια ε, ή ε, έχουν γίνει έχουν ασχοληθεί με τον τουρισμό, τον τουρισμό όπως ονομάζεται ή τον αλλιευτικό τουρισμό σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης. Πρόκειται για γυναίκες οι οποίες ε, ε, ε, διαχειρίζονται όλες τις σχετικές δραστηριότητες με τους άντρες να περιορίζονται στο αλληλευτικό έργο. Ο άξονας 4 ακριβώς αυτό είχε ως σκοπό να υποστηρίξει. Οι γυναίκες αυτές δεν έχουν ε, δεν είναι γεγραμμένες στην κοινωνική ασφάλιση και ε, δεν, το, η εργασία τους ε, δεν υπόκειται σε κάποιο συγκεκριμένο καθεστώς. Βέβαια υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο καθεστώς για αυτές τις γυναίκες με την μεταγραφή της ε, οδηγίας 2010, ε, συγγνώμη, 2010-41 για την ε, ισότητα μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η νέα οδηγία ε, απαιτεί από τα κράτη-μέλη να ανακοινώνουν στην Επιτροπή αν ε, μεταγράφηκε στο Εθνικό Δίκαιο αυτή η οδηγία του 2010. Αυτή τη στιγμή όλα τα κράτη-μέλη έχουν μεταγράψει την οδηγία με εξαίρεση δύο χωρών ε, για τις οποίες έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραβάση ε, και υπάρχουν και τέσσερα κράτη-μέλη τα οποία ε, ζήτησαν παράταση για ορισμένα άρθρα της οδηγίας. Όμως στην πραγματικότητα τελικά η μεταγραφή μιας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο αυτό συνεπάγεται και εφαρμογή της συνεπάγεται ότι η, υφίσταται πλέον ένα ειδικό καθεστώς για τις γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ε, από, για παράδειγμα η Γαλλία από το 1998 διαθέτει τέτοιο κοινωνικό καθεστώς ε, για τις ε, γυναίκες και ε, συντρόφους των αλλιέων. Το 2008 το κοινωνικό αυτό καθεστώς Έγινε υποχρεωτικό ενώ πριν ήταν εθελοντική συμμετοχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ πιο γρήγορη τα τελευταία πέντε χρόνια, από το 2008 και μετά. Δεν λέω ότι η Γαλλία είναι το παράδειγμα, γιατί σε άλλες χώρες υπάρχουν άλλοι τρόποι. Για παράδειγμα στην Πορτογαλία οι γυναίκες δηλώνονται ε, ως εργαζόμενες στα σκάφη χωρίς αμοιβή. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να είναι καλοί μέσα από την κοινωνική ασφάλιση, να έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση, στην επιμόρφωση, στις επαγγελματικές οργανώσεις κλπ. Γιατί μόνο αν δηλώνονται στην κοινωνική ασφάλιση ε, μπορούν οι σύζυγοι και οι σύντροφοι να, αλλιέων να μπουν να γίνουν μέλη επαγγελματικών οργανώσεων αλλιών. Αυτό το ζητούσαν οι ίδιες οι γυναίκες ε, από παλιά σε όλες τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την Ελλάδα, την Ιταλία κλπ. Τώρα, κάποιες συστάσεις. Πρέπει να γίνει υποχρεωτικό, υποχρεωτική συλλογή ε, στοιχείων απασχόλησης ε, με κατανομή φίλο. Είναι ε, πραγματικά κρίμα που δεν έχουμε τέτοιου στατιστικά στοιχεία σήμερα το 2013. Γιατί ε, έχουμε απουσία στοιχείων όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για τους άντρες. Για παράδειγμα, τι εκπαίδευση έχουν οι, οι άντρες. Δεν το ξέρουμε. Πώς θα σχεδιάσουμε πολιτικές όταν δεν γνωρίζουμε σε ποιους απευθυνόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν τα στατιστικά αυτά στοιχεία να είναι υποχρεωτικά και για τους τρεις υποτομείς. Αλία, ε, χθιοκαλλιέργεια και μεταποίηση. Και γιατί να μην ανοίξουμε αυτά τα στοιχεία και στις συντρόφους συνεργάτηδες. Η Γαλλία διαθέτει τέτοια στοιχεία για παράδειγμα αρκεί να τα ζητήσουμε. Που ίσως να θέλουν να τα δίνουν ακόμα και αν δεν είναι και πλήρη. Τρίτο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε στην έκθεση αυτή, την οποία σας καλώ να διαβάσετε, είναι η οργανώση των γυναικών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε δύο τύπους οργανώσεων. Έχουμε οργανώσεις γυναικών αλλιέων, όχι σε όλες τις χώρες, γιατί σε ορισμένες χώρες αυτές οι ε, γυναίκες ε, βρίσκονται, δεν έχουν δικές τους οργανώσεις, είναι σύνδεσες οργανώσεις με τους άντρες, όπως στη Γαλλία για παράδειγμα. Αλλά έχουμε οργανώσει γυναικών, αλλιών, στη Γαλλικία, για παράδειγμα. Και μια άλλη σειρά οργανώσεων ε, γυναικών ή συντρόφων ε, ιδιοκτητών σκαφών και βέβαια πληρωμάτων. Γιατί πολύ συχνά τα ξεχνάμε τα πληρώματα. Αυτές οι ομάδες ζητούν πρόσβαση στην διαδικασία λήψη αποφάσεων, ζητούν κοινωνική ασφάλιση, όπως είπα και προηγουμένως, και τα αιτήματα αυτά σημαίνουν αναγνώριση της συμμετοχής τους στον τομέα της αλίας. Οι σύντροφοι των αλίων και των ηχθειοκαλλιεργητών ε, ε, ε, έχουν οργανωθεί σε ανεξάρτητες οργανώσεις ε, οι οποίες ζητούν και μάχονται για την ισότητα και για την αναγνώρισή τους και προσπαθούν να προωθήσουν την παρουσία των γυναικών και να αυξήσουν και την αμοιβαία τους γνώση μέσω ανταλλαγών μεταξύ τους. Οι γυναίκες, για παράδειγμα, στην ε, Γαλλικία κινούνται χέρι-χέρι με τους ουρανούς των ανδρών, αλλά έχουν ε, μια σχετική άγνοια διαχείριση αυτών των οργανώσεων Εμείς το βλέπουμε αυτό στην καθημερινή επαφή μαζί τους. Ε, υπάρχει επίσης έλλειψη ανανέωσης των ηγετικών μορφών και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε μια όθηση. Και βέβαια η πιο μεγάλη έλλειψη είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Σε ορισμένε χώρε αυτέ οι οργανώσει που είναι τοπικέ οργανώσει έχουν μεγαλύτερο προπολογισμό γιατί οι τοπικές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές τις χρηματοδοτούν, αλλά όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε στο εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, τόσο μειώνεται ο προπολογισμό. Γι' αυτό το λόγο οι γυναίκες ζητούν τη δημιουργία δικτύων εδώ και πολλά χρόνια. Τους το υποσχέθηκε και η ε, Επίτροπος στην τελευταία δημόσια κρόση για τις γυναίκες. Τους το υποσχέθηκε και η στρατηγική ισότητας μεταξύ άνδρων και γυναικών. Εκεί υπάρχει στο παράρτημα ένα, μια φράση η οποία ζητά την δημιουργία οικοδόμηση δικτύων. Είναι προφανές ότι τα κράτη τα οποία ε, συνεισφέρουν στο ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας ε, θα πρέπει να την χρηματοδοτήσουν, όμως δεν κάνουν τίποτα. Ακόμα και το Ισπανικό δίκτυο ε, είναι ένα δίκτυο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις οργανώσεις του τομέα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τις οργανώσεις των γυναικών, γιατί οι άνδρες έχουν καπαρώσει κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, αυτό το δίκτυο. Τέταρτο σημείο, ε, κοινή αλληλευτική πολιτική. Υπάρχουν, υπάρχει το δίκτυο ΑΚΤΕΑ από το 2006 και μετά ε, που έχει ασκήσει πιέσει στα ευρωπαϊκά όργανα. Η πράσινη βίβλος για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής όμως δεν κάνει καμία αναφορά στις γυναίκες και αυτό είναι κρίμα. Γιατί γνωρίζουμε, και είναι κρίμα λέω γιατί γνωρίζουμε σήμερα ε, πως τα αλλιευτικά σκάφη ε, τα καταφέρνουν επειδή έχουν ποσοστώσεις. Όμως οι γυναίκες δεν έχουν ε, πρόσβαση σε αυτές τις ποσοστώσεις γιατί, γιατί οι ποσοστώσεις ανήκουν είτε στο σκάφος είτε στον ιδιοκτήτη του. Οι ίδιες οι γυναίκες όμως δεν έχουν πρόσβαση. Άξονας 4 του Ταμείου και Αλίας. Πράγματι εκεί αναφέρει τις γυναίκες. Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία αναφέρονται οι γυναίκες. Θα πρέπει όμως να πάμε λίγο πιο μακριά κοιτώντας την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας, ε, η ενδιάμεση αξιολόγηση ε, του Ταμείου αυτού μας ε, είχε δείξει ότι η συνεισφορά του Ταμείου στις γυναίκες ήταν ουδέτερη, δηλαδή ελάχιστα θετική, σχεδόν τίποτα. Αντίθετα, ο άξονας 4 του Ταμείου Θάλασσης και Αλίας, το, ο οποίος αξιολογείται αυτή τη στιγμή, δεν μας δίνει τα αποτελέσματα του τι έγινε παλιότερα. Ξέρουμε ότι η Farnet, που είναι η οργάνωση που διαχειρίζεται τον άξονα 4 του Ταμείου Αλίας, ε, οργάνωσε εκδηλώσεις, προσπάθησε ε, να εστιάσει τις συζητήσεις στις γυναίκες, αλλά αν δεν συμμετέχουν οι ίδιες οι γυναίκες, αν δεν συμμετέχουν οι οργανώσεις των ε, γυναικών, δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά. Ε, εδώ σας δείχνω ποια είναι η, συνέπεια, ποιες είναι, ποια είναι η συμφορά του Ταμείου Αλίας, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας, μόνο 55 φλακ τοπικές ομάδες δράσης απάντησαν και κυρίως αυτές οι οποίες ε, είναι δραστήριες υπέρ των γυναικών. Βλέπετε ε, ποια είναι, ποιος είναι ο προπολογισμό ε, ανά σχέδιο στην τρίτη στήλη. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες φλάγκ οι οποίες δεν λειτουργούν ακόμα, οπότε δεν μπορούσαν να μας απαντήσουν. Το Ταμείο Θαλασσιαλίας μας δείχνει ότι έχουμε κάτι συγκεκριμένο αυτό στα χέρια μας, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους, ε, να, πετύχουμε αυτό που ονομάζεται gender mainstreaming, την ένταξη δηλαδή των γυναικών σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ αλλά και σε εθνικό επίπεδο, να τους δείξουμε πού είναι οι γυναίκες γιατί κανένας δεν τις βλέπει είναι πράγματι αφανή. Εκτό από την Ισπανία. Είναι η μόνη χώρα η οποία αποδεικνύει πω τι βλέπει τι γυναίκε. Θα πρέπει επίση να επιλέξουμε δείκτε για να αξιολογήσουμε τα διάφορα διαδοτικά ταμεία ε, σε ό,τι αφορά την ισότητα ευκαιριών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το τέλο, να δούμε αν δούλεψε. Θα πρέπει από την αρχή να έχουμε δείκτε στους οποίου θα αξιολογήσουμε στο ενδιάμεσο και στο τέλο για να δούμε ποια είναι η πραγματική, πραγματική επίπτωση των γυναικών. Νομίζω ότι αυτά είχα να πω. Λυπάμαι που ήμουν γρήγοροι και καστές. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πλήρης και θα έλεγα εξαντλητική η παρουσίαση αυτή. Θα δώσω τώρα το λόγο στις πρώτες ομιλήτριες, μάλλον στις τρεις ομιλήτριες που θα ολοκληρώσω το πρώτο πάνελ. Επειδή όμως καθυστερούμε και θέλω να δώσω το λόγο σε όλους όσους θέλουν να κάνουν σχόλια ερωτήσεις, θα σας πιέσω λίγο ε, θα σας παρακαλέσω να είστε σύντομες ε, και έτσι να μείνει χρόνος για να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στην ε, Δόνια Ρώσα Τσαπέλα Πέρεθ στο Τεχνολογικό Κέντρο της Θάλασσας, ΘΕΤΜΑΡ, ένα ίδρυμα στην Ισπανία, είναι επικεφαλής του κοινωνικο-οικονομικού τμήματος και για θέματα αλίας. Κυρία Τσαπέλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δευτρέα Λίας, κυρίες και κύριοι θα εστιάσω πάνω απ' όλα ε, στη δική μας οπτική γωνία ενός ερευνητικού κέντρου και θα σας πω τι έχουμε δει μέχρι τώρα από την εργασία μας με τις γυναίκες. Καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα θετικό μήνυμα. Σίγουρα υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν, αλλά πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια τα οποία εργαζόμαστε για τις γυναίκες βλέπουμε ότι πέρασαν από την αφάνεια στην ορατότητα και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπεράσαμε απλά το να είναι ορατέ οι γυναίκε, αλλά είναι και αξιοζήλευτε. Παραδείγματο χάρη στην περίπτωση τη Γαλλικία στην Ισπανία, οι γυναίκε που συλλέγουν να χάρη στον επαγγελματισμό ε, και στη διαφοροποίηση, ε, αύξησαν και του μισθού του ε, και κατάφεραν μάλιστα να αμείβονται με μεγαλύτερο, μεγαλύτερο μισθό, ημερομίσθη από τους άντρες. Αυτό ίσως είναι η σημαντικότερη πρόοδος που μπορούμε να επισημάνουμε, αλλά πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν για τις γυναίκες στον τομέα αυτό. Είναι βέβαιο όμως ότι ενώ πριν από κάποια χρόνια η γυναίκα μόνο συνέλεγε το προϊόν, να ψάρευε, θέλετε, μόνο και τις αποφάσεις τις λάμβαναν οι άντρες αποκλειστικά. Εκεί ε, όταν συγκαλεί το μία ε, σύσκεψη έρχονταν άντρες. Τώρα έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση και όχι μόνο γιατί οι γυναίκες δείχνουν επιτόπου ε, και στι συντρόφισσές του, αλλά και στον αλληλευτικό κλάδο γενικότερα πώς έχει εξελιχθεί δική του δραστηριότητα και βοηθά και ανταλλαγή απόψεων, αλλά και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων συμμετέχουν οι γυναίκες. Και έχει και πολιτικά αξιώματα. Οι γυναίκες είναι σε γενικές διευθύνσεις, άρα μπορούν να ευαισθητοποιήσουν γενικότερα την κοινή γνώμη κάνει λοιπόν η γυναίκα, ε, ασκεί δραστηριότητες σε όλους τους τομείς παραγωγή, στην χθιοκαλλιέργεια, στη μεταποίηση, στη συλλογή, ε, σε παραδοσιακούς ε, τομείς που εργάζονται δηλαδή παραδοσιακά άντρες όπως στη Γαλλικία. Σήμερα έχουμε γυναίκες προέδρους των συνεταιρισμών των αλληλευτικών. Δηλαδή αρχίζουν οι γυναίκες ε, να κάνουν την παρουσία τους ε, σε ένα αντροκρατούμενο θα έλεγε κανείς ε, τομέα. Επίσης χάρη στην πολιτική διαφοροποίηση ιδρύουν επιχειρήσεις, οι γυναίκες συμμετέχουν στην θαλάσσια διακυβέρνηση, στηρίζουν την ανάπτυξη των παράκτιων κοινωνιών, συμμετέχουν στους εταιρισμού, στα όργανα λήψη αποφάσεων κτλ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις γυναίκες στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Γαλλικία, που μπορεί βέβαια να εξαχθεί αυτό το παράδειγμα σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, γιατί μιλάμε για την ορατότητα ή την αφάνεια στα στατιστικά στοιχεία, είναι ότι όλη αυτή η δουλειά και η εξέλιξη ε, προκύπτει από το, την ανάγκη για αλλαγή. Για τους άντρες δεν χρειαζόταν αλλαγή, ήταν όλο προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες, αλλά για τις γυναίκες χρειαζόταν οι γυναίκες αυτή την αλλαγή, πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν για να είναι επαγγελματίες, να μπορούν να βρουν τη θέση τους, να αναπτύ, να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ε, και την κοινωνική και την οικονομική των περιοχών τους. Γι' αυτό λοιπόν ε, συμμετείχαν σε δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ήταν οι πρώτες που έδειξαν ότι είναι διτεθειμένες να μάθουν. Ε, ήταν ανοιχτές στη διαφοροποίηση, δημιούργησαν ισχυρές οργανώσεις και έχουν βέβαια πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα και αντοχή. Και όλα αυτά βοήθησαν τις γυναίκες να αναπτύξουν δραστηριότητες ε, εργασίας στο δίκτυο, σε διαδικτύωση δηλαδή. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, ακούσατε και από τους προλαλήσαντες. Πρώτα απ' όλα, μεγάλη, μεγάλο ποσοστό ε, γυναικών ε, απασχολούνται στη συλλογή οστράκων. 3.500 είναι οι γυναίκες, 475 οι άνδρες. Και στην Ισπανία ε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παρουσία, ε, σχεδόν ένα προς ένα ή ίσως και παραπάνω σε κάποιους τομείς ε, είναι οι γυναίκες. Υπάρχουν επίσης γυναίκες που έχουν πτυχία πανεπιστημιακά και μπορούν ε, να είναι ένα μέλη πληρώματος ε, σε ένα λευτικό. Όταν όμως ε, οι πλειοκτήτες αναζητούν προσωπικό προτιμούν άντρες για να πάρουν στο πλήρωμα των σκαφών τους και όχι οι γυναίκες. Εκεί πρέπει λοιπόν να υπάρξει βελτίωση. Επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι οι γυναίκες που εργάζονται στην ηχθειοκαλλιέργεια και θέλω να το τονίσω. Είναι πολύ περισσότερες 20.000 είναι οι άντρες, πάνω από 45.000 είναι οι γυναίκες, αλλά αυτές ε, που έχουν ικανότητες ε, τεχνικές ε, περισσότερες είναι, γνώσεις είναι οι γυναίκες, 530 σε σχέση με 300 τόσους άντρες. Τώρα, για την ορατότητα, για να είναι πιο ορατές οι γυναίκες, είχαμε τη στήριξη της διοίκηση σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό τοπικό επίπεδο και την άμεση υποστήριξη υπαλλήλων που ήταν επιτόπου για να βοηθήσουν τις γυναίκες να οργανωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματισμό μέσω δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, ανταλλαγής εμπειριών και άλλων που αναφέρθηκαν και στην αρχή. Οι γυναίκες αφού δουν πώς οι συντρόφισσες τους, άλλες γυναίκες από άλλες περιοχές, από άλλες χώρες αναπτύσσονται, εξελίσσονται και στον τομέα εργασίας, θέλουν και αυτές να συμμετάσχουν να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και συμμετείχαν γυναίκες σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά project, από το Interreg, στο Equal, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας, τις πρωτοβουλίες. Και πολύ σημαντική έγινε η διαδικτύωση. Στην περίπτωση της Γαλλικίας, οι γυναίκες που ξεκίνησαν, όπως οι συλλεκτρίες Οστράκων, με αυτή τη διαδικτύωση, ε, κατάφεραν να προσελκύσουν, με χάρη τις επιδιορθώτριες δικτυών, που κατάλαβαν ότι και αυτές πρέπει να ε, οργανωθούν. Αυτό μεταφέρθηκε στη Βόρεια Ισπανία, στην, ε, στην Καταβρία, στη Γαλλικία ή στην Πορτογαλία. Υπήρξε και εκεί διαδικτύωση. Στην Ισπανία το Ισπανικό κράτος στηρίζει και ένα Ισπανικό δίκτυο γυναικών στην Αλία για να έχουν προβολή ορατότητα οι γυναίκες. Και αυτό δημιούργησε ντόμινο. Είχε πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα προσέλκυσε, ε, υπήρξε μετάδοση, μεταδόθηκε αν θέλετε το μικρόβιο αυτό της διαδικτύωσης. Και θα ήθελα να πω και για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας ότι διαδραμάτισε και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο τομέα αυτό της ορατότητας, ιδίως με την διαφοροποίηση. Υπήρχαν πολλά project ε, ειδικό που θα μιλήσει για το Φαρνέτ θα σας τα πει πιο αναλυτικά. Εγώ θα ήθελα για τη δική μου περιφέρεια την Γαλλική, να σας αναφέρω δύο ε, project τα οποία χρηματοδότησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Για να δείτε τι αλλαγή έζησαν, βίωσαν οι γυναίκες στον κόσμο της Αλίας. Ε, για, τις, ε, για την περιοχή του Αγγιόλισε, οι γυναίκες που συλλέγουν όστρακα, που ήθελαν να έχουν μεγαλύτερη προστέμινη αξία για τα προϊόντα τους, ήθελαν διαφοροποίηση, όχι απλά να αλλιεύουν, ήθελαν να κάνουν και άλλες δραστηριότητες. Ανέλησαν λοιπόν, λοιπόν και επένδυσαν τα χρήματα και την προσπάθειά τους ε, σε όλη την αλυσίδα αξίας ε, του προϊόντος. Επένδυσαν λοιπόν σε ένα, μια ε, μονάδα για τον καθαρισμό, έκαναν γαστρονομικά εργαστήρια για την εστίαση, τα ξενοδοχεία λοιπά για να βλέπουν όλοι ότι το το προϊόν τους είναι πολύ καλής ποιότητας, άρχισαν να πόλουν απευθείας, πήγαν σε σχολεία για να εξηγήσουν ε, σε τι σύνδεσε τη δουλειά τους, που είναι μια αξιοπρεπής δουλειά που γίνεται από επαγγελματίε πραγματικά ε, και έπειτα βλέπουμε ε, στο πάνω πλαίσιο πώς αυτή η καμπύλη τιμιών του προϊόντος αυτού, του της μεθύστρας δηλαδή, ε, πώς ε, δείχνει ακριβώς αυτή την προστιθέμενη αξία. Η μέση τιμή είναι γύρω στα 5 ευρώ στη Γαλλικία ε, αλλά φτάνει στη δική του κοινότητα στα 9 το κιλό. 9 ευρώ το κιλό. Πολύ θετικό στοιχείο αυτό και δεν εντοπίστε μόνο στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν πολλέ άλλε περιοχέ, όχι Αγιόλς μόνο, αλλά και άλλε περιοχέ. Βέβαια υπάρχουν και περιοχέ με προβλήματα ακόμα. Ένα άλλο παράδειγμα που ήθελα να σα δώσω, που το ξέρει και η Κομισιόν, το ξέρει και το Κοινοβούλιο, είναι το project από μια ομάδα γυναικών από τη Μπαγιώνα που ασχολούνται με τη συλλογή των ε, ε, χινόμιδων περθέμπες τα λέμε στη Γαλλικία. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες ε, συλλέγουν ε, αυτό το προϊόν και το κονσερβοποιούν και έτσι διαφοροποίησαν την δραστηριότητά τους και αύξαν το εισόδημά τους. Ε, δεν συνέλεγαν μόνο λοιπόν τα χινόντα αλλά τα συσκεύαζαν, τα μεταποιούσαν. Και υπάρχουν γυναίκες που δεν προέρχονται από οικογένειες αλλιέων ε, και θέλουν στήριξη αυτές οι γυναίκες. Σε μια συγκεκριμένη μάλιστα ήταν ε, και ε, η πρωτοπόρα για την δημιουργία εταιριών όπως αυτή που λέγεται Μάρντε Σιγέιρο, LTD. Και βλέπουμε ότι σε πολλές οργανώσεις ε, που είχαν επικεφαλής άντρες ε, υπήρξε παρακμή και τελικά ε, διαλύθηκαν, ενώ με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλείας οι οργανώσεις αντίστοιχες με επικεφαλής γυναίκες αναπτύχθηκαν και δημιούργησαν και μια μάρκα που λέγεται 27 Περθεμπέιρας. Ένα σήμα αν θέλετε. Αναπτύχθηκαν λοιπόν. Αυτά είναι τα παραδείγματα που δείχνουν ε, πώς και ε, ο τύπος πλέον να παρουσιάζει ε, τα πράγματα. Αυτό το project το παρουσίασαν ως ένα λαμπρό παράδειγμα στον τύπο. Ως παράδειγμα για τη βιώσιμη αλία. Βέβαια, η λέξη θα δείτε, γρούπο δε ομάδα δηλαδή συλλεκτών ε, οστράκων, στο αρσενικό γράφεται. Εξακολουθεί να γράφεται στο αρσενικό, ενώ θα είναι πιο πολύ θα ήταν καλύτερο να γράφεται στο θηλυκό. Γιατί οι γυναίκες είναι που ασχολούνται. Πραγματική λοιπόν δύναμη ε, που έχουν οι γυναίκες σε αυτό το τομέα. Ε, είναι μοχλός πραγματικά, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα να παρακινήσουν ε, τους συντρόφους και τις συντρόφισσές τους. Έχουν επίσης τη δυνατότητα μεγάλη δημιουργικότητα, να δημιουργούν ιδέες, ε, να είναι επικεφαλής ε, project και έργων ε, με τη συνεργασία και άλλων γυναικών, μεταδοτικότητα επίσης, μετάδοση γνώσεων, διαφοροποίηση. Στα είπα για την αντιπροσώπευση και για την, τα όργανα αποφάσεων. Απλά να πω ποια είναι, ποιες είναι οι προκλήσεις. Πρώτα απ' όλα η ανανέωση, η διαγενειακή, το να μεταφερθεί από τη μια γενιά στην άλλη και να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα επιδόματα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διακρίσεις ακόμη στο χώρο εργασίας, τον ζούμε. Πρέπει λοιπόν να μειωθούν, διαφοροποίηση το είπαμε, αναγνώριση και στην νομοθεσία, να υπάρξει νομικό καθεστώς δηλαδή. Επίσης να βρεθεί ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και προσωπικής ε, οικογενικής ζωής είναι κάτι που μας αφορά όλους. Συνεργαζόμαστε να λέτε όχι, αλλά πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι γυναίκες είναι αυτές που έχουν και τους δύο ρόλους ε, και μεγαλύτερη, καλύτερη εκπροσώπηση, αντιπροσώπηση στα όργανα λήψη αποφάσεων. Σήμερα ο ρόλος ε, της γυναίκας είναι ορατός παντού, υπάρχει τάση να δοθεί μεγαλύτερη αξία και προβολή στη γυναίκα ε, που μπορεί να βελτιώσει την οικονομία. Ακόμη και στο Βατικανό γίνεται λόγος για μεγαλύτερο ρόλο και συμμετοχή των γυναικών Να συνεχίσουμε επίσης ε, να επενδύουμε στην εκπαίδευση των γυναικών, ανταλλαγή εμπειριών ε, σε workshop, ε, εργαστήρια, σεμινάρια για την γαλάζια ανάπτυξη, το είπε και η Διευθύντρια για την ανάπτυξη των ακτών, ναυτιλιακή θάλασσα πολιτική κτλ. κτλ. Και τα συμβουλευτικά, γνωμοδοτικά, λευτικά συμβούλια και ό,τι άλλο όργανο υπάρχει πρέπει να το προωθήσουμε. Έχουμε ένα συμβουλευτικό, γνωμοδοτικό μάλλον λευτικό ε, συμβούλιο στην ε, Γαλλικία που έχει οκτώ μέλη γυναίκες που συμμετέχουν ενεργά. Επίσης, να δώσουμε καλύτερη ε, συμμετοχή συνέχεια και στον Ευρωπαϊκό Ταμείο και νέες ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση μελλοντικές προοπτικές. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα μάλα το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις ε, διαδικτυώσεις, για τις, ε, τις συνεργασίες, συνέργειες ε, και με ερευνητικά κέντρα και ολοκληρώνω όταν μία συλλέκτρια από την Γαλλικία τη ρώτησαν γιατί συμμετείχε ε, στον τέταρτο άξονα είπε ότι όταν κάποιος έχει στόχο, έχει ένα όνειρο, θέλει να το πραγματοποιήσει Δεν μπορεί να σταματάει, πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται, να εξελίσσεται και ε, περιμένεις να βγει ένα νέο πρόγραμμα για να καταθέσεις ε, τις δικές σου προτάσεις. Και κατάφερα πετύχει θαύματα συγκεκριμένη να βελτιώσει την αξιο την προβολή του επαγγέλματό τη και να αυξήσει τα εισοδήματά τη μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Καταρσίνα Βυσόκα από την αλληλευτική κοινότητα της Ούστκα στην Πολωνία. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε σε αυτήν την πολύ σημαντική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει να κάνει με το ρόλο των γυναικών στην αλληλεία μαζί με το σύζυγό μου. Ε, είμαστε ιδιοκτήτες ε, τα τελευταία 17 χρόνια αλλιευτικού σκάφους ε, το οποίο κληρονόμησε ο, πατέρας μου, ο σύζυγός μου από τον πατέρα του. Όσον αφορά το ρόλο των γυναικών στην αλληλεία, στο πλαίσιο της κοινή αλληλευτικής πολιτικής θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η, ότι η αλληλεία υπάρχει μόνο όσο υπάρχουν ακόμα ψάρια. Και ο ρόλος των γυναικών σε αυτόν τον σημαντικό τομέα της ε, οικονομίας έχει ιδιαίτερη σημασία. Ωστόσο, η μεταρρύθμιση της αλληλείας ε, στην Βαλτική ε, κρίθηκε αποτυχία. Είναι μια κλειστή θάλασσα και σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Θαλάσσης πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα. Γι' αυτό οι αλείς της ε, Βαλτικής αντιμετωπίζουν ε, μια καταστροφική κατάσταση. Άλλωστε αυτή η πολιτική στόχο είχε να προστατεύσει τα ψάρια στο οικοσύστημα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να θίξω θέματα που σχετίζονται με την ε, μεταρρύθμιση της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, διότι μέχρι στιγμής η προσέγγιση στα θέματα της Βαλτικής έχει οδηγήσει σε καταστροφική κατάσταση από πολιτιστικής ε, και οικονομικής πλευράς. Ένας Πολωνός Αλιέας ήδη έχει μιλήσει εδώ για την ζημιά που έχει προκαλέσει η βιομηχανική αλληλεία είπε ότι η συνέχιση της αλίας σε βιομηχανικής κλίμακας θα οδηγήσει σε καταστροφή του οικοσυστήματος της Βαλτικής. Κανείς δεν ήθελε να τον ακούσει τότε ε, και τώρα βλέπουμε ότι ο γάδος ε, στη Βαλτική μικραίνει ε, συνεχώς, χάνει βάρος και μπορούμε να το αποδείξουμε. Έχει καταστραφεί η αλία στη Βαλτική λόγω της υπερβολικής αλίας βιομηχανικής κλίμακας και αυτό ε, σημαίνει ότι οι γάβοι δεν βρίσκουν αρκετή τροφή και ε, δεν αναπτύσσονται αρκετά. Η Κομισιόν θέλει τώρα να καλύψει τα λάθη που έχουν γίνει σε συνεργασία με τα λόμπι, τις διάφορες ομάδες ε, ειδικών συμφερόντων. Αποτέλεσμα είναι οι ιδιαίτερα αρνητικέ συνέπειες οι οποίες θα επηρεάσουν όλες τις πτυχές φυσικές και οικονομικές της αλίας. Θα είναι κάτι που θα επηρεάσει τα, ε, ε, τα ψάρια, τα πουλιά και τα θηλαστικά. Οι αλίες ε, χρησιμοποιούν μη επιλεκτικά εργαλεία αλληλείας ε, και δεν ε, ελέγχουν ε, ποσοτικά ή ποιοτικά τα αλλιεύματα. Η Κομισιόν έχει ρυθμίσει τα πάντα στη Βαλτική συμπεριλαμβανομένου του ε, χρώματος των σημαίων, ακόμα και πιο σημαντικά θέματα. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η κοινή αλλιευτική πολιτική έχει οδηγήσει στην καταστροφή αυτή. Υπάρχουν ε, πολλά παραδείγματα κακής διαχείρισης από πλευράς της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όσον αφορά την αλληλεία στη Βαλτική. Θα ήθελα να αναφέρω τον κανονισμό 169 κάθετος 2008. Κάποια είδη εξαιρούνται της ε, υποχρέωσης ε, υποβολής αναφοράς, το οποίο σημαίνει ότι, το, ότι δεν ε, φαίνεται ο συνολικός όγκος των αλλιευμάτων στις στατιστικές. Επίσης, οι λοβιίστες της αλίας βιομηχανικής κλίμακας έχουν καταφέρει ε, να χρησιμοποιούνται ε, δανέζικα σκάφη γρηγρή, ε, κάτι που έχει οδηγήσει σε πολύ σημαντική μείωση του γάδου σημαντικό ποσοστό των ε, αλλιέων ε, στη Βαλτική είναι γυναίκες και λόγω της ε, ανεξέλεγκτης αλλιείας των πελαγικών ειδών που αποτελούν τροφή για τον γάδο, λόγω λοιπόν της υπεραλίευσης αποφασίστηκε να ε, δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα για να ε, σωθεί ο γάδος, κάτι όμως το οποίο τελικά αποτέλεσε αποτυχία. Ε, στηρίχθηκαν νορβηγικές ηχθειοκαλλιέργειες αντί να εφαρμοστούν πραγματικά προγράμματα για να σωθεί ο γάδος. Η Ευρωπαϊκή Αλληλεία βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. μπορούμε να ρωτήσουμε τους ε, υπουργούς ε, στα κράτη-μέλη ε, σχετικά με τα επίπεδα αλληλείας. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να μην βλέπουν πραγματικά το τι συμβαίνει αποφασίστηκε για το 2014 να αυξηθεί κατά 59% η αληθική ε, προσπάθεια. Ε, αυτό λοιπόν αποτελεί ε, παράδειγμα τέτοιας κακής διαχείρισης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης είναι ένοχο στην κακή αυτή διαχείριση. Ε, υπάρχει έκθεση που ε, κρίνει ε, ισορροπημένη και κατάλληλη την προσέγγιση αυτή. Τι θα πούν οι άνθρωποι αυτοί όμως στους αλλοίς και θα ήθελα να σας καλέσω να αντιμετωπίσετε με σοβαρότητα την καταστροφική κατάσταση στη Βαλτική. Η βιομηχανική αλληλεία στην Βαλτική θα οδηγήσει σε εξαφάνιση των ε, ηχθείων και η αλλιευτική προσπάθεια για τα απελακικά είδη θα πρέπει να μειωθεί. Ελπίζουμε αρμόδιος φορέας ε, να εξετάσει την ε, καταστροφική αυτή κατάσταση και να μπορέσει να δει ποιοι είναι ένοχοι για την κατάσταση αυτή. Υπάρχουν προσπάθειες να συγκαλυφθεί η κατάσταση. Σύντομα όμω όλοι οι αλληλεί στη Βαλτική αλλά και από άλλε ευρωπαϊκέ χώρες ε, θα μιλούν για το θέμα αυτό. Ε, στις 11 και 12 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Παρίσι μεταξύ αλλιέων που χρησιμοποιούν επιλεκτικά εργαλεία αλληλείας. Η συνάντηση αυτή στόχο είχε να οδηγήσει σε δημιουργία μιας Διεθνού Ένωση ε, αλλιέων μικρή κλίμακας. Ελπίζουμε ότι η νέα αλλιευτική πολιτική θα αποτελέσει πραγματική μεταρρύθμιση. Μέχρι στιγμής όλες οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν έχουν οδηγήσει σε μείωση της τροφής για τον ευρωπαϊκό γάδο και ελπίζουμε αυτό που ε, συμβαίνει τώρα να αλλάξει στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ε, όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στη Βαλτική. Ε, δυστυχώς ε, δεν ακούσαμε πολλά για τις γυναίκες, πιο πολύ για τη Βαλτική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, οι δύο επιτροπές μας είναι οι πιο αρμόδιες επιτροπές, πώς δεχόμαστε τα σχόλιά σας. Δίνω το λόγο τώρα στην Μπάρμπαρα Ρόντεμπουργκ Κερτσέμα ε, στο Βάντενσε, στο Βάντενσε των κάτω χωρών. Παρακαλώ. Okay, thank Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε σήμερα τη δυνατότητα να μιλήσω εδώ. Εγώ θα ήθελα να θέσω το ερώτημα γιατί οι γυναίκες δεν είναι ορατές στον τομέα της αλληλείας. Όσον αφορά τις κάτω χώρες, αληθεύει ότι οι τομείς της αλληλείας όπου εργάζονται γυναίκες είναι λιγότερο ε, ορατοί. Ε, μιλάμε για την ε, αλληλεία μικρής κλίμακας όπου γυναίκες και άντρες συνεργάζονται και πάνω στα σκάφη και στη στεριά. αλλά αυτοί οι τομείς ε, της αλληλείας έχουν σχεδόν εξαφανιστεί στις κάτω ε, και είναι πολύ λίγο γνωστοί εκτός των κάτω χωρών. Θα σας δείξω κάποιες εικόνες. Βλέπετε εδώ αλληλεία με απλά διακτής. με το οποίο ε, αλλιεύουν ψάρια. Βλέπετε εδώ πέρα μία ε, εικόνα ε, με έναν αλιέα που πιάνει μεθύστρες με λόγχη τύπου σκούπας. Εδώ βλέπετε γρίπο και τα δίκτυα αυτά δεν είναι σταθεροποιημένα, επιπλέον ελεύθερα. Και αυτό σημαίνει ε, ότι ε, τα δίχτυα αυτά μαζεύονται με τρόπο διαφορετικό από τα άλλα. Και εδώ βλέπετε μια εικόνα ε, ηχθιοπαγίδας. Αυτή είναι πολύ παλιά μορφή αλίας Παλαιότερα είχαμε στα ύδατά μας ε, πολύ ε, εκτεταμένη αλληλεία τέτοιου τύπου, αλλά λόγω των φραγμάτων που δημιουργήθηκαν έχει σχεδόν εξαφανιστεί αυτού του τύπου η αλληλεία. Εδώ βλέπετε μία εικόνα από τη Βόρεια Θάλασσα, όπου αλλιεύεται λαβράκι με καλάμι. Ο αλλιέας αυτός ε, πουλάει στην ε, αγορά τα ψάρια του και εδώ βλέπετε εμένα ενώ μαζεύω στρίδια. Όλες αυτές οι δραστηριότητες ε, αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και έχω πολύ κατανόηση για την κυρία από την Πολωνία που μόλις πήρε το λόγο και που επέστησε την προσοχή μας στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλία γενικά. Διότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αλληλείς είναι τα ίδια που αντιμετωπίζουν οι αλληλείς γενικά. Οι κύριες ε, απειλές ε, για την αλία μικρή κλίμακα είναι η καταστροφή των οικοσυστημάτων και των αλλιευμάτων λόγω της ε, ρήπανση, ε, λόγω της ε, ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, στι κάτω χώρε λόγω των φραγμάτων που έχουν δημιουργηθεί, το οποίο σημαίνει ότι έχει έχουν κατακαιρματιστεί τα ύδατα, χρησιμοποιούνται και αντλίες, αλλά και λόγω της κακής διαχείρισης. Και αυτό σχετίζεται σε κάποιο βαθμό Ε, με την εξαφάνιση των παλιών ε, κανόνων ε, σχετικά με το πώς θα έπρεπε να πραγματοποιείται η αλληλεία. Βλέπουμε όμως και την είσοδο αλλιέων από άλλες περιοχές που δεν σέβονται απαραίτητα τις παραδοσιακές κοινότητες αλλιέων. Επίσης αντιμετωπίζουμε την απώλεια της πρόσβασης σε ε, ε, παραδοσιακές περιοχές ε, αλληλείας, ιδιαίτερα στην πόρια Θάλασσα, διότι εδώ συχνά η αλληλεία πραγματοποιόταν σε πολύ ρηχές περιοχές και είναι μια καταπληκτική περιοχή αυτή από πλευράς φυσικής, πολλά σπάνια είδη πουλιών υπάρχουν εδώ για παράδειγμα, αλλά Οι περιοχές αυτές συχνά γίνονται αντικείμενο απαγόρευσης επειδή είναι πολύ σημαντικές περιοχές για ε, τη διατήρηση κάποιων ε, πτηνών. Πραγματοποιούνται και άλλες ε, δραστηριότητες όπως είναι για παράδειγμα η αλληλεία οστράκων, κάτι που επίσης επηρεάζει την αλία και επίσης λόγω των διαφόρων αδειών και ποσοστώσεων. Ε, τελικά ε, οι άνθρωποι των παραδοσιακών αυτών ε, κοινοτήτων αλλιέων χάνουν τα δικαιώματα πρόσβασης επειδή οι άδειες καταλήγουν σε αλλιείς απ' έξω. Έτσι λοιπόν χάνονται αυτά τα δικαιώματα και τελικά τα αποκτούν ε, άνθρωποι από πιο πλούσιες περιοχές ε, που μπορούν να πληρώσουν ε, για να πάρουν τις άδειε. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες σημαίνουν ότι συχνά νιώθουμε ότι είμαστε εμείς ένα είδος υποεξαφάνιση. Πολύ συχνά λοιπόν βλέπουμε ότι οι φώκες, πολλά είδη πτηνών, τα πάνε μια χαρά αναπτύσσονται, αλλά ένας τομέας που επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια είναι η αλληλεία και οι αλληλευτικές κοινότητες ε, απειλούνται. Στην δύσκολη λοιπόν αυτή κατάσταση δεν ξέρουμε πόσο θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Οι γυναίκες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όχι μόνο επειδή συνεργαζόμαστε με τους συζύγους μας και τους συντρόφους μας στην αλληλεία και στο σπίτι και κατά την επεξεργασία και ε, την μεταποίηση και πώληση των ηχθείων, αλλά και επειδή οι γυναίκες νιώθουν ιδιαίτερη ευθύνη για την διατήρηση καλού κλίματος μέσα στην οικογένεια και γι' αυτό επενδύουν πολύ χρόνο και προσπάθεια ε, στο να ενθαρρύνουν ε, τους ε, ανθρώπους και να τους δίνουν ελπίδα. Οι άντρες επικεντρώνονται περισσότερο στα προβλήματα και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και συνεχώς προσπαθούν να συνεχίσουν τις αλληλευτικές δραστηριότητες παρά τις δυσκολίες. Αλλά οι γυναίκες πολύ συχνά, από ό,τι βλέπω εγώ γύρω μου, προσπαθούν να βλέπουν πέρα από τα προβλήματα, προσπαθούν να βλέπουν νέους ορίζοντες, να σκέφτονται νέες εξελίξεις, νέες ε, ευκαιρίες. Και το βλέπω αυτό στις επαφές μου με τους ανθρώπους από αλλιευτικές κοινότητες. Μία από τις ιδέες είναι να είναι πολύ σύντομη η αλυσίδα ε, ε, ε παροχής τροφίμων, διότι έτσι δημιουργείται πολύ θετική ενέργεια και εμείς ε, ως αλληλείς θα γίνουμε πιο ορατοί. Δεν είναι κάτι λοιπόν μόνο που ε, φέρνει περισσότερο εισόδημα, είναι πολύ καλό και για το ηθικό και τα ψάρια που πολλούνται είναι υψηλής ποιότητας. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε αρχίσει να, να πολλούμε ψάρια στο κέντρο του Άμστερνταμ που είναι και το κέντρο της εξουσίας. Ε, κάθε εβδομάδα λοιπόν ε, πηγαίνουμε από, την, από το βόρειο μας των κατοχωρών στο Άμστερνταμ για να πουλήσουμε τα ψάρια μας ώστε ο κόσμος να γνωρίσει και να εκτιμήσει τα προϊόντα μας. Κάτι ε, που θα έχει θετικές επιπτώσεις και σε εμά. Ε, τους λέμε δηλαδή ότι είμαστε εμείς αυτοί που πιάσαμε αυτά τα ψάρια. Ε, πολλές ιδέες λοιπόν προέρχονται από τις γυναίκες και αυτός ο ρόλος ε, επικοινωνίας ε, είναι ένας τομέας όπου οι γυναίκες μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Bien. Finalizado esta primera parte. Τελειώνουμε αυτό το πρώτο τμήμα και θα ήθελα να σας προτείνω, αν συμφωνείτε, ε, αντί να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων στο τέλος κάθε τμήματος, να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή στο τέλος μόνο. Ας ακούσουμε όλους τους καλεσμένους μας και μετά περνάμε στις ερωταποκρίσεις. Νομίζω ότι το θέμα το επιτρέπει. Αν συμφωνείτε λοιπόν, ας περάσουμε στην επόμενη ολυμήτρια, ε, πρόοδος στα προγράμματα ε, ε, του Ταμείου Αλίας. Θα δώσω το λόγο στη Μόνικα Μπουρκ από το δίκτυο υποστήριξης Farnet, ε, του δίκτυου υποστήριξης του άξονα 4 του Ταμείου Αλίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να τελειώσουμε και όλα στην ώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι όσο δυνατό πιο γρήγορη. Θα μιλήσω για τον άξονα 4 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας. Το ΦΑΡΝΕΤ είναι ο φορέας που υποστηρίζει την υλοποίηση του άξονα 4. Να πούμε ποιος είναι ο άξονας 4. Νομίζω ότι ακούσαμε αρκετά σήμερα για αυτόν τον άξονα, καθώς επίσης για τη συνεισφορά του στη, σε ό,τι αφορά την δραστηριότητα των γυναικών. Να σας πω λοιπόν τι είναι ο άξονας 4 και να σας δώσω και μερικά παραδείγματα συγκεκριμένων project ε, έργων που υλοποιούνται. Καταρχήν λοιπόν τι είναι ο άξονας 4. Πρώτα ε, για μια εδαφική προσέγγιση ε, που έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει κλαδικά προβλήματα αλλά και εδαφικά προβλήματα. Ε, για πρώτη φορά έχουμε αυτόν τον άξονα κατά τη διάρκεια αυτής της προγραμματικής περίοδου. Βλέπετε ποια είναι τα προβλήματα. Ε, πολλά από αυτά αφορούν το τομέα της αλίας. Έχουν σχέση με τους ε, φυσικούς πόρους, με την οργάνωση του τομέα, την κατάρτιση, το κόστος των καυσίμων κλπ. Ο... Η λογική είναι η προσέγγιση μας να είναι από κάτω προς τα πάνω μέσω τοπικών ομάδων δράσης ε, και εδώ θέλω να υπογραμμίσω τον ρόλο των γυναικών στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος και ως σύνδεσμος ανάμεσα στον τομέα και την κοινότητα όπως το είπε και συνάδελφος από την Ολλανδία όσο και ε, άτομα τα οποία θα ξεκινήσουν δραστηριότητες διαφοροποίησης και εντός τομέα και εκτός τομέα. Λοιπόν, ο άξονας αυτός υλοποιείται από flags, από ομάδες τοπικής δράσης με στόχο ε, μια συγκεκριμένη περιοχή και με μια συγκεκριμένη στρατηγική ε, που διαρθρώνεται γύρω από μια συγκεκριμένη εταιρική σχέση, μια partnership το, οι αποφάσεις λαμβάνονται τοπικά για το ποια προγράμματα θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Γίνεται εταιρική σχέση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Και όταν μιλάμε για τα προβλήματα του τομέα της αλίας που μπορεί να είναι ίδια για άντρες και γυναίκες, αλλά μπορεί να μην είναι και ίδια, μπορεί να είναι και πιο συγκεκριμένα για τις γυναίκες. Ε, οπότε πρέπει να ληφθούν κάποιε συγκεκριμένε αποφάσεις για το πώς θα δαπανηθούν τα συγκεκριμένα κονδύλια. Αυτές λοιπόν οι ομάδες τοπικής δράσης FLAX θα πρέπει να βοηθούν ώστε να κινητοποιηθεί ο κόσμος σε τοπικό επίπεδο και να στηριχθεί η πρόθεση και η ανάπτυξη τοπικών project. Νωρίτερα είδαμε, τα είπε κάτι φραγκούδι, από τη, για τη μελέτη αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπουμε το 50% των διευθυντών φλάγκ είναι γυναίκες, καλή αρχή είναι αυτή, το 22% των οργάνων που λαμβάνουν αποφάσεις τα φλάγκ είναι γυναίκες. Χαμηλή παρουσία γενικότερα στον ελεκτικό τομέα, το 29% των στρατηγικών έχουν ε, στο επίκεντρό του τις γυναίκες και 19% των project που χρηματοδοτούνται έχουν ε, μία δικαιούχο ή στόχο, ε, κοινό στόχο γυναίκα. Δεν θέλω να διαβάσω ποια είναι τώρα τα επιλέξιμα μέτρα. Υπάρχει μια, ένα ευρύ φάσμα ε, μέτρων που μπορούν να στηρίζονται ανάλογα με το τι θεωρεί η τοπική ομάδα σημαντικότερο. Έχουμε ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ε, της αλληλευτικής περιοχής γενικότερα. Ε, έχουμε αύξηση της προσθέμενης αξίας, συνεργασίες, δικτύωση, οργάνωση ομάδων γυναικών. Όλα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον άξονα 4. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 300 ομάδες τοπικής δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε 21 διαφορετικές ε, χώρες με μέσο όρο 3 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια όλης τη προγραμματικής περίοδου. Βέβαια αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα, από κάτω από 1 εκατομμύριο σε ορισμένε χώρε, μέχρι ε, και 17 εκατομμύρια αν δείτε τα διάφορα, τις διάφορες ομάδες τοπικής δράσης. Τώρα αυτά ήταν η θεωρία. Να δούμε λίγο και την πράξη με παραδείγματα για το τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Βέβαια είναι νωρί ακόμα. Είναι η πρώτη πραγματική περίοδος, ε, όπως ε, σας είπα, για αυτό τον άξονα 4, αλλά ήδη βλέπουμε αριθμό έργων τα οποία έχουν ξεκινήσει. Έχουμε τρεις διαφορετικές ομάδες, οργάνωση και δικτύωση γυναίκων στον αριθμικό τομέα, κατάρτιση των γυναικών και τέλος ε, άμεση χρηματοδότηση η οποία πολύ συχνά λείπει στις δραστηριότητε των γυναικών στο Μετσαλίας. Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ε, ένα οριζόντιο θέμα είναι η υποστήριξη στην ανάπτυξη του project, την υλοποίηση του project. Ε, αφορά και τις τρεις προηγούμενες ομάδες γιατί πολλές, πολύ συχνά οι γυναίκες δεν έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ε, επιχειρηματικά σχέδια κλπ. Οπότε τις βοηθάμε. Τώρα, για την οργάνωση και δικτύωση καταρχήν, στον τομέα της αλίας, υποστηρίζουμε ενώσεις και δίκτυα γυναικών ως ε, πλατφόρμες ε, παρουσίας των γυναικών για την ανταλλαγή εμπειριών. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, έχουμε μια σειρά ε, τοπικών ενώσεων συζύγων ε, αλλιών που δημιουργήθηκαν στην Ανταλουσία. Αυτό δεν υπήρχε, τουλάχιστον όχι σε αυτό το βαθμό. Στην Γαλλικία ναι, υπήρχαν τέτοιου είδου ενό στην Ανταλουσία όχι όμως. Εμπνεύστηκαν λοιπόν από το θέμα της δικτύωσης μέσω της ε, επαφής με άλλες ε, περιοχές και δημιούργησαν και αυτοί τις δικές τους ενώσεις. Και πάλι στην Ανταλουσία έχουμε ένα δίκτυο Συνεργασία ε, μεταξύ των 7 ομάδων τοπικής δράσης Ανταλουσία για τη δημιουργία ενός δικτύου, Ανταλουσιανού δικτύου ε, ενθάρρυνσης των γυναικών στον τομέα τη Αλία να ξεκινήσουν καινούριε επιχειρήσει και εταιρείε. Η ανεργία στην Ισπανία είναι μεγάλο πρόβλημα, οπότε το δίκτυο υποστηρίζει γυναίκες ε, και μέσω μικρών βίντεο αν διηγούνται οι γυναίκες στην εμπειρία με την έναρξη μιας καινούριας επιχείρησης, μιας δραστηριότητα έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν και άλλες γυναίκες ε, και να υπάρξει ένα πολλαπλασιαστικό φαινόμενο. Σε αυτές τις εκδηλώσεις ε, επίσης ε, πολύ συχνά είναι δύσκολο κανείς να συμμετάσχει γιατί πρέπει να ταξιδέψει, να μείνει στη Μαδρίτη, στο Σαντιάγο Δε Κομποστέλα. Οπότε και αυτά χρηματοδοτούνται. Το Φάρνετ άλλωστε και πριν από δύο χρόνια είχε χρηματοδοτήσει την ε, παρουσία ε, ενός αριθμού γυναικών σε ένα μια εκδήλωση που είχε διοργανωθεί στις Βρυξέλλες πριν από δύο χρόνια. Επίσης ε, χρηματοδοτούμε τη βελτίωση των προσόντων μέσω δικτύων, όπως αυτό το δίκτυο της Γαλλικίας. Μετά, σε ό,τι αφορά την επιμόρφωση, ε, είδαμε διάφορα μαθήματα, μερικά ειδικά για γυναίκες, ε, πληροφορική, για συλλογής μαλακίων στη Γαλλικία, επιδιόρθωση δικτύων, ε, χειρισμός των εχθείων και μεταποίησή τους, management και διοίκηση, ε, ακόμα και ε, δραστηριότητες δημιουργίας δερμάτων από, από δέρμα ψαριών στη Φιλανδία και τη Γαλλία. Καταρχήν στη Φιλανδία οι Γάλλοι μετά είδανε το project αυτό, εμπνεύστηκαν, ζήλεψαν και έγινε μια ανταλλαγή τεχνογνωσίας έτσι ώστε να ε, αναπτυχθεί το, η αντίστοιχη δραστηριότητα και στη Γαλλία, όπως και έγινε ήδη. Μετά, άμεση χρηματοδότηση οικονομικών δραστηριοτήτων, για παράδειγμα για την, ε, και για τη βελτίωση του, της ποιότητας ζωής, χρηματοδοτούμε ε, βελτίωση των ασιακών συνθήκων, φροντίδα παιδιών, περιβαλλοντικά σχέδια. Έχουμε υποστηρίξει ε, επίσης την αγορά εξοπλισμού για να βελτιωθεί η εργασιακή διαδικασία, για παράδειγμα μηχανές διαχωρισμού, μαλακίων, ε, μεταφοράς, μικρά, όχι, μικρά σκάφη μεταφοράς ε, αλακτήρια, ε, αποδητήρια μάλλον για, τους, για συλλέκτες μαλακίων, ε, κέντρα επιμόρφωσης, ε, μια αντένα κεραία Wi-Fi για, ε, το, για τα λευτικά σκάφη έτσι ώστε το πλήρωμα να μπορεί να είναι σε επαφή με την οικογένειά του όσο είναι στη θάλασσα, καντίνες, πρόσβαση στο ίντερνετ για γυναίκες και για οικογένειες αλλιέων κλπ. Και βέβαια υπηρεσίε φροντίδας παιδιών όσο οι γυναίκες βρίσκονται στη θάλασσα. Τέλος, η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων. Εδώ περιλαμβάνουμε μερικά πράγματα που είδαμε ήδη προηγουμένως για την βελτίωση του, της προσθέμενης αξίας ε, των τοπικών προϊόντων, διαφοροποίηση, ε, σε καινούριου κλάδους κλπ. Ε, η Ρώσα Τζαπέλα ε, μας, μίλησε για τις συλλέκτες μαλακίων στην Αλιόνς, στον ποταμό Αλιόνς μάλλον. Προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε νέους τρόπους διάθεσης στην αγορά, πρόθεση των τοπικών προϊόντων, χρηματοδοτούμε δραστηριότητες όπως εκδηλώσεις γευσηγνωσίας, ε, δημιουργία νέων μεταποιημένων προϊόντων κλπ. Πολύ συχνά οι γυναίκες ε, προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με άλλους κλάδους, με άλλους τομείς έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν καλύτερα τα προϊόντα τους. Έχουν υποστηρίξει τη μεταποίηση. Η... Πολύ σχετική με τις γυναίκες πάντοτε. Και μετά έχουμε και δραστηριότητε που ξεφεύγουν από τον ελευτικό τομέα. Πάμε στην διαφοροποίηση. Ε, για παράδειγμα ανακαίνιση ενός ελευτικού σκάφους για τουριστικούς σκοπούς, ε, δημιουργία μικρών ξενοδοχείων ή αστιατορίων, ε, οικογένειες οι οποίες μετατρέπουν, μετασκευάζουν το οικογενειακό του σπίτι σε εστιατόριο όπου δουλεύουν οι γυναίκες πολύ συχνά, ε, μια δεύτερη δηλαδή εμπορική δραστηριότητα ή ακόμα και το χρηματοδοτήσαμε και ένα μαγαζί που πουλούσε παγωτά ε, για την κόρη ενός αλία. Επειδή ακριβώς η ανεργία είναι πολύ μεγάλη, ο αλίας, ε, συγγνώμη, η χρηματοδότηση επέτρεψε σε αυτό το κορίτσι να ε, διαφοροποιηθεί τελείως από τον τομέα της αλίας. Τελειώνω με τα συμπεράσματά μου. Οι γυναίκες για μας είναι πρωτοπόρες ε, στην καινοτομία, στην διαφοροποίηση. Ο άξονας 4 επιτρέπει να δημιουργηθούν ε, ενώσεις γυναικών, ε, να βελτιώσουν την οργάνωση και την ορατότητά τους, να συμμετάσχουν σε γυναίκες σε αποφάσεις, στη λήψη αποφάσεων. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή τους στις ομάδες τοπικής δράσης ε, και στα συμβούλια των ομάδων αυτών, γιατί εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις και με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται και η πρόσβασή του στη χρηματοδότηση ε, και για τις υπάρχουσες δραστηριότητες και για νέες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο τρίτο πάντελ, απλά θα σας πω ότι μας μένει μισή ώρα μόνο και για να ολοκληρώσουμε και για να κάνουμε τη συζήτηση. Θα δώσω τώρα την προεδρία στον συνάδελφο Μικαλ Γκούσταυσον για να προεδρεύσει τη ε, συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπατε ακριβώς, ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Παρακαλώ λοιπόν τους υπόλοιπους ομιλητές να το σκεφτούν αυτό. Ε, μάλλον δεν θα έχουμε πολλή ώρα για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ε, θα πρέπει να κλείσουμε στις 6.30 ε, διότι η καταπληκτική διερμηνής μας, λέει ο Πρόεδρος, θα πρέπει να αποχωρήσουν. Δεν θα έχουμε διερμηνία δηλαδή μετά. Δίνω λοιπόν τώρα τον λόγο στην κυρία Ρόζα Σταράς Φεραγκούτ. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πολύ που μπορώ να μιλήσω σε όλους σας για το πολύ αυτό ενδιαφέρον ζήτημα των δικτύων των γυναικών και των ενώσεων στον τομέα της αλίας. Πρώτα απ' όλα κάποιες σκέψεις πάρα πολύ γρήγορα και θα προσπαθήσω να συντομεύσω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρώτη σκέψη, η αφάνεια. Αυτό που το ακούσαμε πολλές φορές σήμερα, ότι πολλές φορές το έργο των γυναικών που, είναι, που εργάζονται στον τομέα της απασχόλησης είναι αφανές. Ε, για την παγκόσμια κατάσταση υγείας και της εκθεοκαλλιέργειας, παγκόσμια κλίμακα για το 2008 σύμφωνα με τη ΦΑΟ, ε, περίπου 48 εκατομμύρια συμμετείχαν στον αλευτικό, το πρωτογενή αλευτικό τομέα άμεσα ή έμεσα ε, και το 12% εξ αυτών ήταν γυναίκες. Ωστόσο, δεν έχουν ληφθεί υπόψη γυναίκες που δεν το δηλώνουν το επάγγελμα, μόνο αυτές οι οποίες ε, πληρώνουν εισφορές και αφορούσε μόνο το ορατό, τις ορατές εργαζόμενες και βέβαια υπάρχουν πολλές άλλες γυναίκες, μητέρες, ε, σύζυγοι, κόρες ε, που εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις και που κάνουν όπως το είπαν και πολλοί ε, προλαλήσαντες, πολλαπλά καθήκοντα και μέσα στην αιστεία και εκτός και με την κοινωνική ζωή ασχολούνται και σχεδόν πάντοτε αναλαμβάνουν πλήρως ε, και τις ε, σχέσεις με την τράπεζα, με τη διοίκηση, ε, με τις επαγγελματικέ οργανώσεις και ούτω καθεξής ως συνεργάτηδες του ΑΛΕΑ αυτό που θεωρώ ότι είναι πρώτα πολύ σημαντικό είναι να γίνουν ορατές οι γυναίκες αυτές. Και το πρώτο πρόβλημα είναι ότι παραμένουν αφανείς ή παρέμεναν αφανείς ε, μέχρι πολύ πρόσφατα. Δεν είχαν καμία αναγνώριση όπως είπαμε. Πάντως αρχίζει να βελτιώνεται αυτή η κατάσταση. Είχαμε την οδηγία 86-613, τροποποιήθηκε από την 41 οδηγία του Ευρωκοινοβουλίου με στόχο ακριβώς να έχουμε ορατότητα για τον τομέα αυτό, να θεσπιστεί ένα νομικό καθεστώς, ώστε οι σε αυτές να έχουν πρόσβαση ε, στις κοινωνικές παροχές, προνοιακά επιδόματα, διαμετώρητες κτλ. Ε, και βέβαια να παίρνουν σύνταξη και να έχουν και επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της αλίας. Επίσης ε, εισάγεται και όρος ε, του συντρόφου νόμιμου, συμβιούντο, συμβιούντος που δικαιούται επίσης να έχει τέτοιου είδους παροχές. Σε δύο κράτη, Αυστρία και Ρουμανία, κινηθεί η διαδικασία παράβαση. Τα άλλα έχουν εφαρμόσει τα σχετικά μέτρα. Βλέποντα τώρα τα στατιστικά στοιχεία, λείπουν δείκτε για να δούμε ακριβώ ε, πόσε γυναίκε εργάζονται στη μεταποίηση ή στην ηχθειοκαλλιέργεια και υπάρχουν πολλές διαφορές ε, μεταξύ κρατών μελών όπου η γενική απασχόληση στην Ιρλανδία για παράδειγμα είναι κάτω από το 30% ενώ στην Πολωνία πάνω από το 60%. Όπως και να έχει πάντως το σίγουρο είναι ότι καλό θα ήταν να υπάρχουν αξιόπιστοι δείκτες για να έχουμε αξιόπιστα δεδομένα σε καθέναν από τους τομείς γιατί τα στατιστικά στοιχεία ε, που έχουμε και ο μόνος τρόπος για να πάρουμε στοιχεία για την αλληλεία είναι μέσω μιας κοινή ανάλυση ε, των ε, στοιχείων που δίνουν οι τρεις τομείς, αχθιοκαλλιέργεια, αλληλεία και μεταπίση. Δεν έχουμε στοιχεία μόνο για τον κάθε τομέα δηλαδή. Επίση, η συγκέντρωση στοιχείων που γίνεται, η συμπίληση στοιχείων και τροποποίηση που γίνονται είναι σημαντικέ για να έχουμε αυτού του δείκτε. Τελευταία μου σκέψη είναι ε, σε σχέση με τις γενικές οργανώσεις. Νομίζουμε ότι είναι τεράστια η σημασία τους. Μπορούν να είναι πάρα πολύ σημαντικοί συνομιλητές και σημαντικός μοχλός για την επίτευξη όλων αυτών που θέλουμε. Στην ε, Νορβηγία και στην Ιρλανδία ξεκίνησαν αυτές οι γενικές οργανώσεις ε, και κινητοποιούνται στις κοινωνικές πτυχές ε, της άλλης βελτίωσης συνθήκων εργασίας, βελτίωση της επικοινωνίας των ανδρών που είναι πάνω στο σκάφος και των οικογενειών του στη Στεριά. Βέβαια, από την δεκαετία του 80 και μετά δημιουργήθηκε ένας Είχαμε πολλαπλασιασμό τέτοιων οργανώσεων Έχουμε επίσης ε, πολλές διεκδικήσεις που σχετίζονται πάντα με την επιβίωση αυτού του τομέα στην αρχή και μετά ε, στην ε, περάσπιση, στην προάσπιση μάλλον του στόχου για την δημιουργία νομικού καθεστώτος. Ακούσαμε τις γενικές οργανώσεις, μιλήσαμε για αυτό το ίδρυμα στη Γαλλικία και για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Είδαμε λοιπόν πως αυτές οι οργανώσεις με νύχια και με δότια προασπίζονται τις προκλήσεις αυτές που έχουν αντιμετωπίσουν οι γυναίκες και ότι έχουν ε, όλες αυτές τις δυνατότητες για να πετύχουν πολλά και πετυχαίνουν ε, πολλά. Για τη Γαλλική συγκεκριμένα και τη χώρα των Βάσκων, οι οργανώσεις αυτές είναι πάρα πολύ δυνατές ε, στην Ισπανία και θέλησαν να, να δώσουν επαγγελματικό χαρακτήρα σε αυτές τις δραστηριότητες που ήταν άτυπες μέχρι τότε. Οργάνωσαν λοιπόν μαθήματα εκπαίδευσης και βέβαια ό,τι άλλη δράση είναι απαραίτητη για, την, για το μεγαλύτερο επαγγελματισμό. Είπαμε για την ακτέα ε, που είναι και ευρωπαϊκή εκπρόσωπος αν θέλετε αυτών των οργανώσεων. Επίση, να πω ότι πολλέ μικρέ κυρίω και τοπικέ οργανώσει αντιμετώπισαν προβλήματα χρηματοδότηση για να μπορέσουν να επιβιώσουν, ιδίω αυτή την κρίση που βιώνουμε. Αλλά νομίζω ότι με την ακρόαση αυτή φαίνεται πια ότι οι οργανώσει αυτέ, αν επιβιώνουν, επιβιώνουν γιατί είναι σημαντικέ για την επίτευξη των στόχων που αναφέραμε όλοι εδώ και πιστεύω μας βρίσκουν όλους σύμφωνους. Τέλος, θέλω να τονίσω το ρόλο των γυναικών στην κοινή ελευτική πολιτική. Θα γνωρίζετε ότι για τα ταμεία συνοχή, τα μία ταμεία, κάποια θέματα έχουν κλείσει, κάποια όχι. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας, έχουμε το Ταμείο για την Αλία και τη Θάλασσα και ένα από τα θέματα που συζητούνται ακόμα ε, είναι τα εκ των προτέρων, δηλαδή ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών και αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να είναι κάποιος επίδοξος δικαιούχος των κονδυλίων αυτών των ταμείων. Ένα άλλο κριτήριο είναι η ισότητα ευκαιριών για άτομα με αναπηρία και στην προκειμένη περίπτωση γυναίκες με αναπηρία. Και αυτό είναι ένα εγκάρσο άξονα και άλλους εξάντε όρο, εξάντε εκ των προτέρων δηλαδή, προϋπόθεση να μην υπάρχει διακριτική μεταχείριση σε γυναίκε με αναπηρία, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια των ταμείων. Έτσι θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το ρόλο των γυναικών στην κοινή λευτική πολιτική. Και εδώ ολοκληρώνω ευχαριστώντα για μια ακόμη φορά την Επιτροπή Αλίας και την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών για το ανακρόαση αυτή και όλου όσου ε, παρενέβησαν μέχρι τώρα στη συζήτηση. Eh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θίξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο σχετίζεται με την έλλειψη ορατότητας. Ε, δυστυχώς, οι γυναίκες δεν είναι αόρατες εντό αγωγικών μόνο στον τομέα της αλληλείας, αλλά σε, πολλά, σε πολλούς τομείς. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε παντού στην πατριαρχική κοινωνία μας. Όπως και να έχει προχωράμε, στον επόμενο ομιλητή, στην επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Κριστίν ε, Εσκαγέ. Ε, σας δίνω το λόγο, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, εδώ και χρόνια ε, μελετώ την εξέλιξη των αλευτικών κοινοτήτων στην Πορτογαλία και τις πορτογαλόφωνες χώρες και παρακολούθησα την αλλαγή που έγινε με την ένταξη της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1986. Η πολιτική της χώρας ήταν να επενδύσει στις, ε, ε, στα λιμάνια πέντε φορές περισσότερο από ό,τι στον υπόλοιπο τομέα. Ε, οι, οι δομές έγιναν πιο σύγχρονες, έγιναν πιο αυτόματες και αυτό δημιούργησε σε, οδήγησε σε αλλαγή των δραστηριοτήτων με μείωση των γυναικών και μετατροπή των δραστηριοτήτων σε τουριστικές. Εδώ θα δείτε τον πίνακα αυτό με την μετακίνηση σε άλλες δραστηριότητες. Για παράδειγμα αυτό είναι η πόλη του Ναζαρέ... της Ναζαρέ στην Πορτογαλία. Αριστερά βλέπετε τις δραστηριότητες ε, και μετά της Αλίας το 1986 και με μετά το 1986, αριστερά πριν το 1986, δηλαδή στη μέση του πίνακα, βλέπετε ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες γινόντουσαν από γυναίκες. Μετά το 1986 βλέπετε ότι είναι από άντρε. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα για την Ισπανία, την Ελλάδα, την Γαλλία κλπ. Χώρες οι οποίες συμμετέχουν, συμμετείχαν στο πρόγραμμα γυναίκες στην Αλληλεία και στην ηθιοκαλλιέργεια στην Ευρώπη που ονομάζεται πρόγραμμα FAM. Είναι ένα θεματικό δίκτυο ε, που χρηματοδοτήθηκε από το τέταρτο πρόγραμμα πλαίσιο. Γνωρίζουμε ότι στις περισσότερες αλληλευτικές κοινότητες ο ρόλος των γυναικών ε, είναι κρίσιμος, παρόλο που δεν αναγνωρίζεται συχνά. Όταν έφτασα στη Μαδέρα το 1997, ε, δεν είδα απλώς αφάνεια των γυναικών, είδα την απουσία των γυναικών, την εξαφάνιση των γυναικών. Πλην όμως τα στατιστικά του 2011 ε, έδειχναν 25 αλληλείς γυναίκες, ζητώ συγγνώμη, λέει ομιλήτρια, και ε, μία ιδιοκτήτρια σκάφους. Αλλά ε, τόσο στο λιμεναρχείο όσο και στα τοπικά αρχεία κανείς δεν μπορούσε να τις εντοπίσει, ούτε να πει καν το όνομά τους. Σε ό,τι διαφορά τις Αζόρες ε, αλληλείς και γυναίκες αλλοιών υπάρχουν ακόμα. Ε, που είναι γυναίκες ε, Αλλά για πόσο χρόνο ακόμα. Η κατάσταση στα πορτογαλικά αρχιπελάγια είναι πραγματικά ανησυχητική όπως μας ε, δείχνει αυτή η συγκριτική ε, μελέτη αζωρών και μαδέρας. Βλέπετε πόσο μειώνεται ο, α, ο πληθυσμός ε, και βλέπετε ε, και πόσο ε, έχει αλλάξει ο αριθμός των οικογενειακών, των μελών της οικογένειας που εργάζονται χωρίς να αμείβονται. Σε ό,τι διαφορά τις ενώσεις, οκτώ ενώσεις στις Αζόρες, εκ των οποίων τρεις είναι γυναικών. Στη Μαδέρα η μόνη ένωση που υπάρχει αναφέρει ότι ένα μέλος της μόνο είναι γυναίκα αλλά την εκπροσωπεί ο άντρα τη. Δηλαδή η ίδια δεν συμμετέχει ποτέ στι συνεδριάσει. Στην Μαδέρα, στον τομέα τη Αλία δεν υπάρχει καμία ένωση γυναικών. Ε, δεν υπάρχει βασικά ούτε ένωση καν πλεξίματος, πλεκτριών ε, στην Μαδέρα σε ό,τι αφορά τι γυναίκε. Αλλά ε, είτε μιλάμε για την Πορτογαλία είτε για άλλε χώρε οι γυναίκε αυτέ αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και όλες αναρωτιούνται για το μέλλον των ενώσεών τους και το μέλλον τους μέσα στην Ευρώπη. Ως απάντηση σε αυτή την ανησυχία το πρόγραμμα FAM δημιούργησε το ε, δίκτυο ακτέα, ευρωπαϊκό δίκτυο ακτέα, του οποίου ένας στόχος ήταν να τις ε, βοηθήσει να είναι περισσότερο παρούσες αυτές και οι ενώσεις τους εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις και για την ηλία και για την ηχθειοκαλλιέργεια. Επίσης να προστατεύσει τα δικαιώματά τους ε, εντός της ε, οικογενειακής επιχείρησης. Ο στόχος του προγράμματος FAM λοιπόν ήταν ε, να δράσουμε υπέρ μιας συλλογικής δράσης των γυναικών με δημιουργία οργανώσεων γυναικών εκεί που δεν υπήρχαν, οργανώσεων γυναικών εκεί δεν υπήρχαν και ε, τη δικτύωση των οργανώσεων αυτών για την ανταλλαγή των πρακτικών. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων. Στον πίνακα υπαριθμών 1 αριστερά θα δείτε ότι το δίκτυο αυτό δημιούργησε ενώσεις γυναικών στην Ελλάδα, την Ιταλία κλπ. κλπ. Ενώ στο δεξιό πίνακα, στο πίνακα αριθμό 2, θα δείτε ε, ε, ότι ενώθηκαν επίσης μια ντουζίνα περίπου ενώσεων. Ε, πλην όμως από το 2010 και μετά ε, δεν βλέπουμε πολύ δραστηριότητα. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να σας δώσω πληροφορίες πιο συγκεκριμένες για το τι απέγιναν. Ποιες είναι, ποια είναι τα συμπεράσματα για σήμερα ε, βλέπουμε μια πολύ μικρή δραστηριότητα αυτών των ενώσεων, συμμετοχή τους σε κάποιες εκδηλώσεις που διοργανώνται από ε, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η σημερινή ακρόαση ε, ή διάφορες άλλες ε, εκδηλώσεις, όμως καμία άλλη δραστηριότητα. Η, η απουσία των ενώσεων, για παράδειγμα των, της Γαλλικίας σήμερα από εδώ, το δείχνει αυτό άλλωστε. Δείχνει ότι υπάρχει προβλήματα κόστους στη μεταφορά. Ε, είναι σημαντικό να τις, να τις στηρίξουμε όχι μόνο μέσω προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα της διαχείρισης οργανώσεων τέτοιου τύπου όταν υπάρχουν, αλλά να τις υποστηρίξουμε και χρηματικά ε, σε ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση των ε, project τους, για παράδειγμα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις νέες οργανώσεις ή τις οργανώσεις επαγγελματικών σωματείων όπως στην Πορτογαλία. Θα Πρέπει να διατηρήσουμε αυτά που έχουν υπάρξει όμως, έχουν δημιουργηθεί ήδη. Ε, οι, όμως οι τέτοιου είδους οργανώσεις χρειάζονται ηγέτη. Εν τω μεταξύ, μέχρι να δημιουργηθούν τέτοιοι ηγέτες, η ακτέα έπαιξε το ρόλο της. Ε, όμως ε, θα πρέπει να δούμε και το μέλλον. Οι ενώσεις αυτές βασίζονται στην εθελοντική εργασία και είναι δύσκολο, δεν έχουν έσοδα, ε, για παράδειγμα να εκδώσουν ένα περιοδικό, μια εφημερίδα. Ε, θα μπορούσαμε να τις βοηθήσουμε σε αυτό ή να τις βοηθήσουμε οργανώνοντας ε, εκδηλώσεις ή συνέδρια στα οποία θα μπορούσαν να βρεθούν μεταξύ τους και να συζητήσουν. Όπως είπε και η Κάτια Φραγκούρη, ε, να σας υπενθυμίσω ότι σε προηγούμενη ακρόαση η Επίτροπος Δαμανάκη είχε ε, δεσμευθεί να βοηθήσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου, αλλά τα τελευταία μισή χρόνια δεν έγινε γίνει τίποτα. Τελειώνοντας να πω ότι θα πρέπει να δώσουμε στις γυναίκες τα μέσα και σε εμά τα μέσα να υλοποιήσουμε τις φιλοδοξίες μας, τις ευρωπαϊκές μας φιλοδοξίες. Και η τελευταία μου σύσταση είναι να μην ξεχάσουμε να διευρύνουμε τις δράσεις μας προς Ανατολάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μας ε, μίλησες για, τις, ε, για τα δίκτυα που υπάρχουν και για τα δίκτυα ενδεχομένω που δεν υπάρχουν, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν. Και περνάμε στην ε, τελευταία ομιλήτρια, την κυρία Ισάουρα Πινιέρο Εσπερών. Ζητώ συγγνώμη για εκεί κακή προφορά μου, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καταρχά, θέλω να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω στη δημοσιευτή ακρόαση. Νομίζω ότι βοηθούν τέτοιες ε, εκδηλώσει για να γίνει καλύτερα γνωστή ως ο ρόλος της ε, γυναίκας ε, στην Ευρώπη και για τη βελτίωση της κατάστασής της. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μπιλμπάο Μπαραντίκα που με προσκάλεσε και γενικότερα για το άνοιγμα στην βασικέ στις βασικές οργανώσεις. Μεγάλο μέρος της ιστορίας χώρας των Βάσκων ε, σχετίζεται με τη θάλασσα. Πολλοί Βάσκοι, πολλές Βάσκες ζουν και ε, εργάζονται στη θάλασσα και για τη θάλασσα την 1η Δεκεμβρίου του 7 οι γυναίκες από το Βόρειο Καταβρικό Πέλαγος ε, συναντηθήκαμε στο δικό μου Δήμο όπου εργάζομαι πάνω από 30 χρόνια στη συσκευασία των ψαριών για να δούμε καλύτερα τι μπορούμε να κάνουμε ε, για έξι χρόνια περίπου ε, οι γυναικές οργανώσεις, οι οργανώσεις γενικά βελτιώσαμε την κατάσταση, δα, λάβαμε βραβεία, αναγνώριση από διάφορους θεσμούς, αλλά σίγουρα ακόμη έχουμε να κάνουμε πολλά για να βελτιώσουμε τις κοινωνικοεργασιακές μας συνθήκες, να αναγνωριστούμε ως κομμάτι ε, του αληφτικού κλάδου. Στη χώρα των Βάσκων έχουμε τρεις οργανώσεις Στην τρίτη των συσκευαστριών είμαι εγώ πρόεδρος. Πρέπει να σας πω ότι είναι μαζί μου εδώ ε, η Μάιτε ε, και η Αϊνόα που είναι οι πρόεδροι των άλλων δύο οργανώσεων, δηλαδή αυτών που εργάζονται για τη συλλογή των ε, ψαριών και για αυτές που εργάζονται για την επιδιόρθωση των δικτύων. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα των Βάσκων, πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Πρώτα απ' όλα οι λεγόμενες νεσκατίγιας εκφορτώτριες. Οι εκφορτώτερες δηλαδή έχουν να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα. Είναι πρώτα απ' όλα γυναίκες, μητέρες ε, ή κόρες των αλλιέων. Όταν φτάσουν αυτοί στο λιμάνι, εκφορτώνουν το σκάφος, πάνε ε, για να πουλήσουν το εμπόρευμα, το πολλούν, επίσης προμηθεύουν και εξοπλίζουν το σκάφος ε, με τα απαραίτητα εφόδια. Ε, για να μπορέσουν οι αλείς έπειτα να βγουν στα ανοιχτά. Είναι ένα ε, επάγγελμα πολύ παλιό μένα, αλλά δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς και επειδή υπάρχει και παροπισμός πολλών σκαφών μένουν χωρίς ε, δουλειά πολλές από αυτές τις γυναίκες. Ε, επίσης έχουμε τις επιδιορθώτριες δικτυών που σε περισσότερες περιπτώσεις είναι πάλι συγγενείς των αλλιέων και επιδιορθώνουν, μπαλώνουν ή φτιάχνουν τα δίκτυα που χρησιμοποιούν ε, τα σκάφη στα λιμάνια μας. Πολλές φορές εργάζονται χωρίς ωράριο, σε κακές καιρικές συνθήκες, με πολύ μικρό και οι μελλοντικές τους ε, προοπτικές δεν είναι καθόλου ελπιδοφόρες. Ε, για τη δουλειά τους απαιτείται πλήρη ετοιμότητα και Πέτυχαν πολλά τα τελευταία χρόνια, ιδίω ό,τι αφορά ε, τις λιμενικές υποδοχές ή τα λιευτικά εργαλεία. Και έπειτα οι συσκευάστριες που υπάρχει μόνο σε ένα λιμάνι όταν φτάνουν και γίνεται η εκφόρτωση των ψαριών, ξεκινούν τη δράση τους οι συσκευάστριες, τα ε, τα, τα ψάρια τα βάζουν ε, σε κασέλες, τα βάζουν πάγο, τα ξυνομούν και με βάση το μέγεθος, ε, ξεκινάνε από το βράδυ μέχρι το πρωί πρέπει να είναι όλα έτοιμα ώστε να ε, μπορέσει το ψάρι να πάει στη νυχτεόσκαλα για πώληση. Ουσιαστικά δουλεύουν μία μέρα τη βδομάδα και το μέλλον τους είναι πολύ αβέβαιο. Αυτές λοιπόν οι τρεις, ε, αυτά τα τρία επαγγέλματα θα έλεγα είναι γυναικεία κατεξοχήν, περιθωριακά σε πολλές περιπτώσεις ε, τα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και είναι αφανή ε, για, τον υπόλοιπο, για τους υπόλοιπους εργαζομένους. Ναι, μεν λοιπόν έχουν γίνει πρόοδοι και γίνονται σε άλλους τόμους, όπως είναι η συλλέκτωση των αμαλακίων. Σε εμά οι συνθήκες εργασίας μας από πάρα πολλά χρόνια μέχρι σήμερα οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει ειδική επαγγελματική κατηγορία ε, μέσα στους επαγγελματίε ε, που εργάζονται στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις. Και επίσης τα έσοδα, τα εισοδήματα είναι πάρα πολύ μικρά. Και βέβαια επειδή ε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαγενειακή ανακύκλωση έχουμε προβλήματα. Άρα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες οι καλές συνθήκες ούτε σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, ούτε σε ό,τι αφορά τις απολαβές. Το ωράριο είναι άτακτο, δεν υπάρχουν Βίωνε μελλοντικές προοπτικές και πρέπει να πω τα τελευταία έξι χρόνια παρόλα αυτά καταφέραμε να πετύχουμε διάφορα. Ιδίω οι συντρόφισές μας ε, που ασχολούνται με την επιδιόρθωση των ε, δικτυών. Ε, καλύτερη εκπαίδευση έχουν, καλύτερη σε εργασιακές συνθήκες, έχουν ενημερωθεί για την πρόληψη, για τα εργατικά ατυχήματα, η διαφοροποίηση. Έχουν πάρει επίσης και ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύει την ειδικότητά του και το ίδιο θέλουμε να επιτύχουμε και τις άλλου δύο κλάδου. Έχουμε ειδική ενδυμασία επίση καταφέρει για να μπορούμε να εργαζόμαστε με μεγαλύτερη άνεση, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμη ζητήματα από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε την 1η Δεκεμβρίου του 6 μέχρι τώρα είναι κάποια που δεν έχουν επιληθεί. Και τι πρέπει να γίνει. Πρώτον, πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα ώστε να υπάρξει αναγνώριση του επαγγέλματό μα ε, και θα πρέπει να προωθηθούν τα επαγγελματικά προσόν. Είπαμε ότι μία κατηγορία, οι επιτευχθόντρες έχουν ε, πάρει το πιστοποιητικό τους, αλλά εμείς θέλουμε το 2013 να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες και για τις άλλες δύο κατηγορίες. Δεύτερον, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι συντελεστές, οι συγκεκριμένοι που ισχύουν γιατί θέλουμε να είναι μικρότερη η ε, ηλικία συνταξιοδότησης γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες εργασίας. Δεν έχουμε όμως ε, προχωρήσει καθόλου σε αυτόν τον τομέα. Καλές προθέσεις, ωραία λόγια, αλλά στην πράξη ουδέν. Τρίτον, αναγνώριση των ε, εργασιακών αναγνώριση επαγγέλματό μα ω βαρέω ενδεχομένω, γιατί δεν αναγνωρίζονται τα αχήματα που παθαίνουμε ω επαγγελματικά. Επίση, κοινωνικο-οικονομικά μέτρα στήριξη ε, πρέπει να τα ε, υιοθετήσουν ε, οι αρχές. Γιατί για διάφορους λόγους εμείς μένουμε ακάλυπτες και μετέωρες. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, κανένα έσοδο, κανένα εισόδημα αν παροπληστεί το σκάφος για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουμε να εισφέρουμε ε, στα διάφορα ταμεία. Ελπίζουμε να είμαστε δικαιούχοι στο Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλία και πραγματικά σας παρακαλώ να συνεργαστείτε μαζί μας για να μπορέσουμε να πετύχουμε πάνω σε αυτό. Θέλω να μας θεωρήσετε και εμάς κομμάτι αυτού του κλάδου, γιατί είμαστε κομμάτι του κλάδου. Επίσης... Por último, έχουμε πρόβλημα με το ότι έρχονται, ε, παρισφρίουν ε, από άλλα επαγγέλματα ε, στο δικό μας το επάγγελμα. Επίσης, για τη χάραξη της αλευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμμετέχουμε και εμείς ενεργά για τη διατύπωση των προτάσεων. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας, γιατί θεωρούμε ότι είναι δίκαιο και σωστό να είμαστε παρούσες στα διάφορα βήματα συζήτησης, δομές όπου συζητείτε και αποφασίζετε το μέλλον του ευρωπαϊκού Αλευτικού τομέα. Πολύ απλά γιατί και εμείς είμαστε ένα κομμάτι, επαναλαμβάνω, του κλάδου και εμείς από πλευρά μας δεσμευόμαστε να εργαστούμε σκληρά για να είμαστε ορατές και στην κοινωνία και στις διάφορες δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις για να βελτιώσουμε τις εργασιακές μας συνθήκες και για να πετύχουμε την αναγνώριση του επαγγέλματός μας. Ολοκληρώνοντας, θα σας πω τη φράση με την οποία κλείσαμε τη διακήρυξη της 1ης ε, Δεκεμβρίου του 2007. Θέλουμε να είμαστε ορατές. Ευχαριστώ πολύ που μας περιγράψατε την ε, κατάσταση στην χώρα των Βάσκων. Καταφέρατε να θίξετε και πολύ σημαντικά θέματα που σχετίζονται με το τι θέλετε να πετύχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγα, λίγα λεπτά μόλις μας δώσανε για πολύ, πολύ σύντομες ερωτήσεις και πολύ, πολύ σύντομες απαντήσεις. Πολύ λίγο χρόνο έχουμε. Το πολύ ένα λεπτό για τις ερωτήσεις. Δύο ή τρεις βουλευτές μπορούν να θέσουν ερωτήσεις και το πολύ μια ερώτηση αναπάντηση. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά γνωρίζετε ότι οι διερμηνεί μα εργάζονται από τις 3 η ώρα, χρειάζεται να κάνουν διάλειμμα, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ. Thank you, Chairman. Well, I... Ο κύριο Άγνιο, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έμαθα κάτι νέο σήμερα ότι ε, υπάρχει πατέ από χινόμυλα ε, και Βρισκόμαστε τρία χρόνια πίσω από την Επιτροπή Άγκρη στο θέμα ε, αυτό, το θέμα των γυναικών δηλαδή. Ε, εμένα με ανησύχησε γενικά το θέμα της γεωργίας και των γυναικών, διότι ε, προκύπτουν πολύ καυτά ερωτήματα. Να σας θυμίσω ότι η Αλία και η Γεωργία ήταν οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Γεωργός είμαι, τρία, τρία αγόρια έχω. Δεν μπορώ να κάνω διακρίσεις ε, στη δουλειά αυτή. Ε, στη Γεωργία βλέπουμε ότι οι γυναίκες ε, τίνουν προς κάποιες, κάποιους συγκεκριμένους τομείς και οι γυναίκες ε, δεν ε, θέλουν να εργάζονται με μηχανές ε, συνήθως, έτσι λοιπόν μπορούμε να τις εξωθήσουμε από τον τομέα. Και όλη αυτή η γραφειοκρατία τελικά θα οδηγήσει σε περισσότερα ψάρια στη θάλασσα, εγώ αμφιβάλλω. Διότι το ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό είναι πολύ κακό και... Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Παρακαλώ, κύριε Σκοπάσικ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι πολύ που ακούω ότι έχουμε μόνο ένα λεπτό για να θέσουμε ερωτήσει μετά από μια τόσο σημαντική ακρόαση. Είναι ουσιαστικά δυνατή η συζήτηση. Ένα συμπέρασμα από μένα, λοιπόν. Έχουμε μια θεωρητική και μια πρακτική προσέγγιση στις γυναίκες στον τομέα της αλληλείας θεωρητικά. Έχουμε ένα τεράστιο πακέτο δυνατοτήτων, πρακτικά όμως η κατάσταση στο, στις κάτω χώρες και στην Πολωνία ε, δεν έχουμε γυναίκες ε, στον τομέα της αλληλείας και οι μικρές ε, και η αλληλεία μικρής κλίμακας ε, υποβαθμίζεται. Δεν ήθελα να θέσω το παράδειγμα αυτό, αλλά όπως ακούσαμε σήμερα, ο ρόλος των γυναικών περιορίζεται ε, στο να έχει κανείς ένα κατάστημα παγωτών. Δύο ερωτήσεις έχω προς την κυρία Ρισότσκα. δεδομένης της κατάστασης ε, στη Βαλτική, ε, πώς βλέπετε το μέλλον των γυναικών στον τομέα της αλληλείας ε, υπό το φως της παρούσας κατάστασης, και έχω και μια ερώτηση προς την κυρία Ρόντεμπουργκ. γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει τόσο μικρό ποσοστό γυναικών στον τομέα αυτών. Κυρία Μπιλμπά Μπαραντίκα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Μάιτε, την κυρία Κόιτε και, τη, και τον Λεάνδρο Άτκο που είναι εδώ μαζί μας σήμερα από τη χώρα των Βάσκων. Τους ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνουν εγώ δεν κατάφερα να είμαι εδώ γιατί χρειάστηκε να είμαι σε άλλη επιτροπή, αλλά ξέρω ότι έγινε λόγος για την ορατότητα και για την αφάνεια. Ε, οι γυναίκες μπορεί να είναι αφανείς, αλλά κάνουν πάρα πολύ κρίσιμη δουλειά στο τομέα της αλίας. Δεν θα υπήρχε ο τομέα της αλλιώς. Θα ήθελα να ρωτήσω την Μόνικα Βούρτς, που αναφέρθηκε σε όλες τις ενισχύσεις που είναι διαθέσιμες. Να τη ρωτήσω αν πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά σωματεία, οι ευρωπαϊκές ενώσεις γνωρίζουν επαρκώς τους, ε, τα μέσα που διατίθενται στην Ευρώπη και αν ε, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ενημερώσουμε όλες τις ενώσεις, τις ευρωπαϊκές ενώσεις ε, για την ύπαρξη της δυνατότητας χρηματοδότησης μέσω αυτών των μηχανισμών. Μετά, σε ό,τι αφορά την ε, παρέμβαση Σάουρα για το τι μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη, εμείς έχουμε υποβάλει πολλές τροπολογίες οι οποίες ε, λήφθησαν υπόψη και στην μεταρρύθμιση και στο Ταμείο, αλλά δεν νομίζω ότι ακούστηκε και πολύ η φωνή μας. Ε, δεν νομίζω ότι το Κοινοβούλιο έδειξε ευαισθησία εναντί των τροπολογιών που υποβάλαμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε. Και όπως είπε ο Σέουρα, ένα κομμάτι της ε, παρεμβασής της αφορούσε τις κοινωνικές φορές και τις τα αιτήματα προς το Υπουργείο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο καθένας από εμά να είναι δραστήριο σε εθνικό επίπεδο. Ο κ. Ρωμέβα, τελευταίος, ε, τελευταία παρέμβαση από Ευρωβουλευτή. Θα ήθελα και εγώ να επωφεληθώ, μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο να γίνει συζήτηση, θα ήθελα να επωφεληθώ για να υπογραμμίσω τα εξή δύο. Πρώτον, το είπαν πολλές ομιλήτριες, ε, θα πρέπει να τελειώνουμε με την αφάνεια. Και όχι μόνο την αφάνεια στις στατιστικές, αλλά και την αφάνεια σε ό,τι αφορά την λήψη ε, συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων ε, το είδαμε ότι υπάρχουν πολλές ενώσεις που χρειάζονται τις βοήθειες αυτές. Ας αναγνωρίσουμε λοιπόν όσα έγιναν μέσω διαφόρων πρωτοβουλειών, αλλά σε νομοθετικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο, δεν έχουν γίνει όλα όσα μπορούσαν να γίνουν. Δεύτερον, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστεί ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, ότι δηλαδή τελικός δικαιούχος θα είναι όλες αυτές οι ενώσεις που αν δεν τις αναφέρουμε ρητά μπορεί να εξαφανιστούν στην πράξη. Νομίζω ότι στην έκθεσή μας, ε, ε, το οποίο το ανέφερε και η Ντολόρες, όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί ήδη. δεν είναι δυνατόν να δώσω το λόγο σε άλλους ομιλητές. Έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Η ε, κυρία Βυσόσκα, η κυρία Ρόντεμπουργκ και η κυρία Μπούς, ε, στις οποίες αναφέρθηκαν οι ομιλητές, μπορούν να πάρουν το λόγο μας. Ευχαριστώ πολύ. Τι να σας πω τώρα. Αν μιλήσουμε για την αλία στην Πολωνία. Σε λίγο δεν θα έχουμε αλία στην Πολωνία. Γιατί, γιατί δεν θα μείνουν ψάρια. Και το λέω γνωρίζοντας τι, τι λέω. Δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα ακόμα αλλά τι έχουμε εκεί, γάδο, σολομό και ρέγγα. Δεν έχουμε και πολλά άλλα είδη. Αν συνεχίσουμε έτσι, ε, πού θα φτάσουμε. Ε, μας προτείνεται ε, διαφοροποίηση, όμως ξέρετε ποιο είναι το κλίμα εκεί πέρα στη Βαλτική, και στην Πολωνία. αν χάσουμε την αλία, καλύτερα να κλείσουμε την πόρτα και να φύγουμε. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Πολύ περισσότερο που δεν θα έχουμε ψάρι ούτε για το δικό μας πληθυσμό. Δεν βλέπω μέλλον για την αλία στην Πολωνία. Μάλλον σε λίγο θα εισάγουμε τα ψάρια μας από την Νορβηγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρόντεμπουργκ. Ευχαριστώ. αν υπάρχουν ε, πολύ λίγες γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό στη θάλασσα, αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές έχουν παιδιά. Οι ναυτικοί ψαράδες φεύγουν για πολύ καιρό από το σπίτι τους, άρα οι γυναίκες θα πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. Και επίσης ε, δεν υπάρχουν μόνο οι ψάρες που λείπουν για πολύ καιρό, αλλά υπάρχει και η μικρή σκλήμακα σαλία που κρατάει μια μέρα το ψάρεμα, το πρωί τέλο πάντων, οπότε οι γυναίκες εκεί απασχολούνται. Υπάρχουν γυναίκες όπου απασχολούνται. Συμφωνώ πάντως με αυτά που είπε η συνάδελφός μου από την Πολωνία. Πρέπει να βρεθούν ε, θέσεις εργασίας. Ε, υπάρχει το θέμα σίγουρα του γάδου. Υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να βρούμε λύσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης το πρόβλημα που υπάρχει με τις για το λαβράκι. Δεν θα πρέπει να πάψει η μικρή κλίμακα παράκτη αλλή, ε, αλλά κοντεύουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Κυρία Μπέρτς. Όσον αφορά την ερώτηση σχετικά με τις ενώσεις γυναικών και το αν γνωρίζουν αρκετά τι οικονομικοί πόροι είναι διαθέσιμη. Είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτό. Ξέρω ότι η Ακτέα γνωρίζει τα θέματα αυτά. Είμαστε σε επαφή μαζί της ε, τα, τα τελευταία χρόνια. Τους προσκαλούμε στις εκδηλώσεις μας σε τακτική βάση. Ε, δημοσιεύουμε τα όσα κάνουν και αντιστρόφως. Το αν όμω όλε οι οργανώσει γυναικών που σχετίζονται με την αλληλεία γνωρίζουν ε, τα θέματα αυτά είναι δύσκολο να το απαντήσουμε. Είναι ο ρόλος των τοπικών ομάδων δράσης ε, να εξηγήσουν στις κοινότητες ότι υπάρχουν ε, αυτοί οι πόροι. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, υπάρχουν πολλά να γίνουν. Απομένουν πολλά να γίνουν ακόμα. Αλλά σε χώρες όπου οι γυναίκες αποτελούν προτεραιότητα, οι τοπικές οργανώσεις, τα φλάξ είναι αρκετά δραστήρια. και προσπαθώντας ε, να ε, πετύχουν περισσότερη συμμετοχή των γυναικών ε, στα Συμβούλια Λήψης Αποφάσεων αλλά και στις επαφές τους με τις ενώσεις γυναικών. ώστε οι γυναίκες να μπορούν να παρουσιάζουν προγραμμάτα στήριξης. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδώ να παίξει σημαντικό ρόλο, στηρίζοντας δίκτυα όπως είναι η ακταία οικονομικά αυτό σίγουρα θα ήταν πολύ χρήσιμο. Τα κράτη-μέλη μπορούν όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ε, των ε, φλαξ να διασφαλίσουν ε, τα θέματα φύλου να αναφέρονται στις στρατηγικές που παρουσιάζουν. Σε κάποιες χώρες οι γυναίκες στην Αλία λένε ότι τα προβλήματα τους είναι ακριβώς τα ίδια με τα προβλήματα των ανδρών και ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται αρκετά καλά στα συμβούλια και δεν νιώθουν δεν θεωρούν ότι είναι θετικό να διαχωρίσουν τους άντρες από τις γυναίκες. όλα εξαρτώνται λοιπόν από τη χώρα. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχουμε χρόνο για τη συζήτηση. Συμφωνώ ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που είναι παρόντες, όλους όσους συμμετείχαν, ε, όλους τους ομιλητές και ευχαριστώ και την Επιτροπή Αλληλείας ε, για τη συνεργασία της. Ε, προσβλέπω και στη συνέχιση της καλής συνεργασίας και ευχαριστώ πολύ και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος, για την απίστευτη υπομονή τους μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ. simplemente reiterar Ευχαριστώ πολύ τον συμπρόεδρο κ. Κωνσταύσον. Ένα πραγματάκι μόνο θέλω να σας να πω. Ε, νομίζω ότι ένα πράγμα έγινε σαφές σήμερα, ότι σήμερα ε, η γυναίκα στην Αλία ήταν λίγο πιο ορατή εδώ μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ.